Right, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν ήδη περάσει οι τρεις, είναι τρεις και έξι λεπτά, γι' αυτό λοιπόν προτείνω να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Καθίστε λοιπόν και ηρεμήστε αν είναι δυνατόν. Ωραία. Σημείο 10 της ημερησία Ο Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 18, όλα τα τμήματα μπορούμε να, κάνουμε, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία απευθεία, εκτό και αν θέλει ο εισηγητή να πει κάτι. Όχι από ό,τι φαίνεται. Επομένω, Κριστιαν, σε ευχαριστούμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα ψηφίσουμε κατά δύο τμήματα, ε, το βλέπετε γιατί έχετε και δύο χωριστούς ε, καταλόγους ψηφοφορίας. Διαδικασία προϋπολογισμού 2018, πρώτη τροπολογία. 5288 ε, υπέρ κατά αποχέσε εγκρίνεται 5269 υπέρ κατά αποχέσε απορρίπτεται 5270 υπέρ κατά αποχέσε απορρίπτεται 5270 ε, συγγνώμη, 52-50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52-27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-09 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52-30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52-31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 52-10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52-51 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο με τις επαληθεύσεις, ηλεκτρονική επαλήθευση, λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας ε, εγκρίνεται. Το επόμενο καταπίπτει, 52 θα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 52-72, ε, απορρίπτεται, 52-73 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 52-74 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 52-75 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 52-28 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 5276 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5319 19 και 53 20 σε μία ψηφοφορία Α, και τις επόμενες τρεις τροπολογίες ε, ψηφίζουμε on block υπέρ, κατά, αποχές 52'77 ε, 52-77 υπέρ, κατά, αποχές 53'15 ε, 53-15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52-78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 52-11 υπέρ, κατα αποχέσε, αποχές εγκρίνεται. 53-12 υπέρ κατα αποχέσε, αποχές εγκρίνεται. 52-79 υπέρ κατα αποχέσε, αποχές απορρίπτεται. 52-61 υπέρ κατα αποχέσε, αποχές απορρίπτεται. 53-16 υπέρ κατα αποχέσε, αποχές εγκρίνεται. 52-62 υπέρ κατά αποχέσε απορριπτεται απορρίπτεται 52-23 υπέρ κατά αποχεσε εγκρινεται εγκρίνεται 52-80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52-81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52-29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52-82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 52-83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 52-12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτη και επομένως block vote 5290 και 5308 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 5284 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5291 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 5291 αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. και εγκρίνεται με σαφή πλειοψηφία. Καταπίπτει η επόμενη 52-26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση, ωραία. Αφού θέλετε, 52-26, ε, τροπολογία Αουστρεβίσιους, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται. τροπολογια 5313, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52-52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πολύ ωραία. Τροπολογία 52-52 σολέ πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. 52-14 καταπίπτει, 52-20 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση από τις 52-20. Άρχεται η ψηφοφορία. Λείπουν τρεις ψήφοι. Δύο, μία ψήφος. Ψήφισαν όλοι. Α, όχι, ο ένας κοιμάται ακόμα. Ε, ωραία. <laughs> Εγκρίνεται λοιπόν με σαφή πλειοψηφία. Επομένως, καταπίπτουν οι δύο επόμενες τροπολογίες και φτάνουμε στην 53-14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52-33 υπέρ. Κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 52-33 άρχεται η ψηφοφορία. Και εγκρίνεται 32 ψήφοι υπέρ 32 κατά. Η επόμενη καταπίπτει 53-18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52-34 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 52-40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52-41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. 52 52-41 ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, σαφώς εγκρίνεται. Σε 52-41 υπέρ, συγγνώμη, 52-15 υπέρ, 52-15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52-22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52-35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Μετά έχουμε ε, ψηφοφορία on block με, για πέντε τροπολογίες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 52-32 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 53-10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53-11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52-94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επίσης. Έχουμε τώρα την ε, συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52-16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 52-55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 52-97 καταπίπτει, 52-98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52-49 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε. Τροπολογία 5249, ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας και ε, κατεψηφίστη. 5302 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5303 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5307 καταπίπτει. Μετά έχουμε ψηφοφορία unblock υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 5360 σολέ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τέλος η 5221 υπέρ κατά αποχές ε, θα ελέγξουμε το αποτέλεσμα ψηφοφορία επί της τροπολογίας 5221 άρχεται Λείπουν τρεις ψήφοι. Πέρα της ψηφοφορίας και σαφέστατα εγκρίνεται η τροπολογία 5221. Τώρα, θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης για τον προϋπολογισμό του 2018. Εισηγητής ο κύριος Πρέντα, συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές ε, θα κάνουμε μια επαλήθευση για την τροπολογία 19 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας 35 υπέρ 30 κατά εγκρίνεται λοιπόν Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές η Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 27 του κυρίου Καστάλντο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 25, Μιχαήλ Γκάλερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 29, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30, υπέρ, κατά, αποχές, Προτιμώ να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική λοιπόν επαλήθευση από τις τροπολογίες 30 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απερίφθη. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται. Ηλεκτρονική λοιπόν τώρα ψηφοφορία επί τροποποιημένου κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε όλες τις ψήφους που χρειαζόμαστε. Εγκρίνεται λοιπόν 49 ψήφοι υπέρ, 12 ψήφοι κατά 5 αποχές. Σας ευχαριστούμε και προχωράμε. Επόμενο θέμα είναι το υπερθμό 11, Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωσης Αφρικής, μια όθηση για την ανάπτυξη. Η συγητής είναι ο κύριος Καστάλντο. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε συγητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους τους συναδέλφους ε, για την εξαιρετική συνεργασία, ε, οι οποίοι λοιπόν παρά την καλοκαιρινή ραστόνη ε, συνεργάστηκαν καλά και επομένως μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα το οποίο μπόρεσε να συμμεριστεί το μεγαλύτερο μέρος της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ για μία ακόμα φορά για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Καστάλντο. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 30. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ή 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα, τροπολογία 5 της κυρίας Βερζιά, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 61 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 34 προς 30. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Την 33 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική εννέα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 7. Βαλέρο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 67 υπέρ κατά αποχές έλεγχος αυτής που είναι η 67. Πέρας. Δεκτή. 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 76 ε, ε, και 79 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έλεγχος, έλεγχος. Ψηφίζουμε την 83, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σχέδιο γνωμοδότης όσο τροποποιήθη υπέρ... Όχι, όχι, ποιος είναι υπέρ. Αυτή είναι ηλεκτρονική, συγγνώμη. Πέρας. Δεκτή. 54 προς 7. Πάμε τώρα στο 12. της, ε, σύναψη συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΛΑΚ. Ο κύριος Περμόη θέλει να πει κάτι. Κυρία Λόζινγκ, ευχαριστώ. Ο Χαβιέ Κούσο Περμούι δεν μπορούσε να έρθει και μου ζήτησε να ζητήσω συγγνώμη και να εκφράσω την λύπη ε, να ευχαριστήσω τους Σκιώδης και την καλή συνεργασία που επιτρέπει την ενδυνάμωση πολιτικού διαλόγου και δημιουργία ενό χώρου για πολιτικές και οικονομικές ανταλλαγές. Ο Χαβιέ Κούσο θέλει να ευχαριστήσει και τα άλλα μέλη που στήριξαν τη συμφωνία, ούτως ώστε να δημιουργηθεί το Ίδρυμα αυτό το οποίο θα βαθύνει τη στρατηγική εταιρική σχέση και θα ενισχύσει και τον διαπεριφερειακό πολιτικό διάλογο. Θα εμβαθύνει τις πολιτικές σχέσεις ώστε να αποκτήσουν την πλήρη τους δυναμική και να ε, δράσουν θετικά απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Και τώρα προχωρούμε στην ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα έχουμε μία τροπολογία του James Carver. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 59 προς 2. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, μα περισσεύει χρόνο από το πρόγραμμα και αυτό είναι θετικό. Α συνεχίσουμε όμω τη συνεδρίαση. Η σύμβολη του ΕΛΚ, παρακαλώ κυρία Όπερμαν, κύριε Όπερμαν. Λοιπόν. Να προχωρήσουμε. Σημείο 13. Ετήσια έκταση σχετικά με την εφαρμογή της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Θα συζητήσουμε λοιπόν την ετήσια αυτή έκθεση. Σας έχει μοιραστεί ένα σχέδιο έκθεσης πριν το καλοκαίρι. Κάποιοι από εσά ελπίζω να είχαν την ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά. Όπως θα ξέρετε, αυτή είναι η πρώτη έκθεση ε, δική μου ε, ως πρόεδρος. Προσπάθησα να επικεντρωθώ στο στρατηγικό σκέλος σε ό,τι αφορά τους στόχους μας, ε, ε καθώς και μια αξιολόγηση του τι συνέβη ε, το περασμένο έτος. Έχετε λάβει και την έκθεση της Αντιπροέδρου της κυρίας Μογκερίνης, είπα της εκπροσώπου για το 2016, οπότε εξετάστε και αυτήν την έκθεση πριν συζητήσουμε το τελικό περιεχόμενο της δικής μας έκθεσης. Έχω εδώ διαρθρώσει την ε, έκθεση με βάση τα τρία ε, βασικά στοιχεία, τους τρεις πυλώνες. Πρώτον, συντονισμός της αξιολόγησης των προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η ενδυνάμωση και η διεύρυνση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και τρίτον, η συνεργασία μέσα σε συμμαχίες και ε, θεσμούς που προωθούν την ασφάλεια. Προσπάθησα λοιπόν να επικεντρωθώ στα πιο σημαντικά ζητήματα. Βεβαίως από εκεί και πέρα εσείς με τις τροπολογίες σας ε, θα μου πείτε τι θεωρείτε εσείς σημαντικό. Εγώ θα σας ενθάρρυνα πάντως να επικεντρωθείτε περισσότερο σε, τομείς και όχι σε γεωγραφικά ζητήματα πιο πολύ σε τομεακά ζητήματα. Λοιπόν, αναμένω τη συνεργασία μας με ανυπομονησία. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα μηνύματα κλειδιά ενώπιση του ερχόμενου έτους, θα έλεγα, να μην υπάρξουν επικαλύψεις με άλλες εκθέσεις. Όπως και πέρυσι, ε, βεβαίως ε, αναμένω τροπολογίες ε, αυτά από την πλευρά μου θα ήθελα τώρα να ακούσω τις δικές σας απόψεις για την έκθεση αυτή. Έχουμε έως τις 5 παρα 20 για το θέμα αυτό, δηλαδή μία ώρα. Βεβαίως μπορούμε να τελειώσουμε και νωρίτερα. Για την ομάδα των Σοσιαλιστικών και Δημοκρατών, ο κύριος Φλάκενστάιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη δουλειά πάνω στην έκθεση και ευχαριστούμε και τον Πολωνό Σύμβουλο, του οποίου την παρέμβαση μπορούμε εδώ και εκεί να δούμε. Δεν έχουμε σοβαρές δυσκολίες με τα λεγόμενα γραφόμενά σας. Σε κάποια σημεία μπορούμε να κάνουμε κάποιες προσθήκες, όπως την κοινή θέση για το εμπόριο όπλων ή να πούμε λίγο περισσότερα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Συμφωνούμε με την στρατηγική συνεργασία με τις ΙΠΑ, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον νέο πρόεδρο για τον οποίο γίνονται καινούριε σκέψεις που πρέπει και αυτέ να τις συμπεριλάβουμε στη δουλειά μας. Σωστά είναι και πολλά από αυτά που γράφεται για τη Ρωσία. Ίσως όμως θα πρέπει να προσθέσουμε μια πρόταση σχετικά με το πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, τι λύσεις θα δοθούν, ε, καταπολέμηση της δημοκρατίας, με ανατολικό και εδώ ενδεχομένως θα πρέπει να γράψουμε κάποια πράγματα. Πάντως η γενική γραμμή της έκθεσης είναι ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό αποδεκτή από εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φλέγκενστάιν. Και τώρα από την ECR ο κύριος Τάνοκ. Όχι. Όχι. Δεν ακούμε τον κύριο Τάνο γιατί είναι εκτό μικροφώνου. Το στείλαμε τον Ιούλιο από ό,τι μου λένε. Έχει κάποιος κάποιο αντίγραφο εδώ. Μπορεί να το διαβάσετε και εν τω μεταξύ να ακούσουμε τον κύριο Νάρτ από την Άλντε, από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ, Ντέιβιντ. Η έκθεση αυτή είναι πολύ καλή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία όμως. Το σημείο 7. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τη φιλοσοφία αυτή να είμαστε στα σύννεφα και να λέμε ότι θα υποστηρίζουμε ε, την κυβέρνηση του Φαγέντ Ελσαρά στη Λιβύη. Πρόκειται για ένα, μια ανύπαρτη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση φάντασμα που δεν ελέγχει καν την Τρίπολη όπου υποτίθεται ότι έχει έδρα. Όλοι οι πρόεδροι, όλες οι κυβερνήσεις ευρωπαϊκές, η Ιταλική, η Γαλλική, η Βρετανική, τελικά αναγνώρισαν ότι ο βασικός άξονας της πραγματικότητας στη Λιβύη είναι εκεί, στη Λιβύη. Δηλαδή, ο Χαλίφα Χάφτερ. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Το να λέμε ότι θα υποστηρίξουμε την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας είναι σαν να υποστηρίζουμε το τίποτα και να κάνουμε πολιτική επιστημονικής φαντασίας ο Υπουργός Εξωτερικών του, του Ηνωμένου Βασιλείου επισκέφθηκε τον Χαλίφα Χάρτερ, τον δέχτηκε και ο Γάλλος υπουργό. Τελικά όλες οι κυβερνήσεις τελικά κάποια στιγμή έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα και όχι με φαντασιακές κυβερνήσεις. Τώρα, το σημείο 20. Θα πρέπει να Το να λέμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία του Μίνσκ, εντάξει. Όμως η συμφωνία του Μίνσκ δεν τηρείται από καμία από τις δύο πλευρές, διότι ούτε και η Ουκρανία έχει τροποποιήσει ε, το σύνταγμά τη για να δεχτεί τον, το αυτόνομο χαρακτήρα μιας περιοχής. Ε, βεβαίως, ε, να βοηθήσουμε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά υπάρχει τεράστια διαφθορά ε, στην παρούσα κυβέρνηση της Ουκρανίας. Δεν μπορούμε, να, δεν μπορούμε να μιλάμε τίποτα γι' αυτό. Όλοι οι υπουργοί που έχουν οριστεί από το εξωτερικό για να υπάρξει μια νομιμότητα και μια αξιοπιστία από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Αμερικανό, τον κύριο Χασέσκο, στον Υπουργό Οικονομίας, που είναι, από, είναι προέλευσης, στον Υπουργό Υγείας, που είναι από τη Γεωργία, ή ο ίδιος ο κυβερνήτης ε, της Οδυσσού, ε, του οποίου του αφαιρέθηκε ε, η εθνικότητα. δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε κυβερνήσεις δια, διαφθαρμένες. Διότι αυτό ζημιώνει την εικόνα μας, την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι τελικά οι πολίτες των χωρών αυτών, της Μολδαβίας ή της Ουκρανίας είναι αυτοί που πλήττονται από τις δια, διαφθαρμένες κυβερνήσεις τις οποίες υποστηρίζουμε εμείς. Και κάτι άλλο τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα έδαφος που λέγεται Ταϊβάν. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ουδετερότητα στη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ταϊβάν, σε ό,τι αφορά τα στενά εκεί. Πρέπει να μιλήσουμε για ειρήνη μεταξύ δύο καθεστώτων οικονομικά διαφορετικών. Είναι μια ζώνη ε, που βρίσκεται σε μεγάλη ένταση λόγω της ε, απειλής Βορείου Κορέας. Πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε και αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νάρτ και τώρα από την Γκουε η Σαμπίνε Λεζινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ για την έκθεση. Από την πλευρά μου η έκθεση πρέπει να πω ότι εστιάζει πολύ στα θέματα ασφάλειας και τις επιπτώσεις θεμάτων ασφαλείας Δηλαδή πάμε προς μια κατεύθυνση εξασφάλισης της ή ε, ασφαλιοποίησης της εξωτερικής πολιτικής. Πολλά θέματα όμως δεν λύνονται μέσα από το πρίσμα της πολιτικής ασφάλειας, αλλά είναι κοινωνικά θέματα και οι στρατιωτικές επεμβάσεις δεν μπορούν να ε, αντιμετωπίσουν τα αίτια των συγκρούσεων. Ε, πολλά από αυτά που λέτε για τα αίτια της ε, φυγής από άλλες χώρες, πρόληψη, αντιαντίδραση, όλα αυτά είναι σωστά. Επίσης ε, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για οδούς νόμιμης μετανάστευσης. Όλα αυτά όμως είναι σε αντίφαση με την τωρινή ενωσιακή πολιτική που βλέπουμε η καγκελάριος να συνεργαστεί με την Αφρική και να ε, θεωρήσει ως ε, δυνατότητα φυγής την δυνατότητα και μόνο ως, ως ε, αίτιο φυγής, τη δυνατότητα φυγής. Ε, δεν μπορεί κανείς να περιοριστεί σε αυτό, θα πρέπει να μπει βαθύτερα στα αίτια που αναγκάζουν τους ανθρώπους να μεταναστεύουν. Τώρα, για την ε, πολιτική προς τη Ρωσία. Παρατηρώ και πάλι ότι είναι σύνθετη η διαμάχη εδώ. Αν δούμε δηλαδή πώς, ε, ποια ήταν η γένεση της κρίσης στην Ουκρανία, το βλέπουμε αυτό. Έτσι λοιπόν, βαθιά αίτια δεν μπορούμε εμείς να τα αντιμετωπίζουμε επιφανειακά και να ε, τα λύνουμε ε, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία. Ε, ούτε βεβαίως θα πρέπει να κραδένουμε ή να ανεχόμαστε ανθρώπους να κραδένουν όπλα. Εμάς η πολιτική μας είναι να προλαμβάνουμε και να αποτρέπουμε τους πολέμους ε, ε, οι βίαιες αντιπαραθέσεις μπορεί να κλιμακώσουν ανεξέλεγκτα την κατάσταση εκεί. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται λοιπόν. Τώρα, για την υποστήριξη των ε, περιφερειών στην Αφρική, παράγραφος 12. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να στηρίξουμε τις αφρικανικές χώρες ώστε να προσανατολιστούν μακροοικονομικά ε, σε ένα θετικό περιβάλλον. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά μου φαίνεται ότι κανείς δεν με... Μιλώ, ε, ε, και δεν μακούτε. ακούτε. Ε, είναι σημαντικό όμως να συζητήσουμε λίγο, να μας... ο, ο παρεμβαίνει ο πρόεδρος και λέει «Έχω πολλά στο κεφάλι μου, αλλά πάντα σας ακούω πολύ προσεκτικά». Ε, εντάξει, ε, αν, αν παρεξήγησα κάτι να με συγχωρείτε. Πάντως επανέρχομαι και λέω, είναι σημαντικό να υπάρξει στήριξη σε ένα συνολικό μακροοικονομικό πλαίσιο. Ε, πάντα μιλάμε για εταιρικέ σχέσεις ε, δημοσίου ιδιωτικού τομέα της ΔΙΤ. Ε, δεν τα όλα αυτές οι συμπράξεις. Ε, οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνονται σε δημόσιους τομείς όπως σε εκπαίδευση, υγεία, σε συνεργασία με εταίρους από την κοινωνία των πολιτών. Και θα πρέπει να σταματήσει η μονόπλευρη εμπορική πολιτική προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα για την ε, παγκόσμια στρατηγική της Ένωσης, ε, εδώ υπάρχουν ορισμένες ε, διαφορές μεταξύ μας. Δεν θέλουμε στενότερη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Επίσης, απορρίπτουμε αυτό το αίτημα το 2% του ΑΕΠ να επενδύεται στο στρατιωτικό τομέα. Ε, δεν θέλουμε ε, προγράμματα για την στρατιωτικοποίηση της ΚΕΠΑ. Ε, εδώ υπάρχουν διαφορές προς, την, προς το σχέδιο έκθεσης λοιπόν. Γι' αυτό θα καταθέσουμε μια έκθεση μειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ συνάδελφες, σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε λέει ο κύριος Μέζεριξ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την έκθεση. Είναι μια καλά διαστρωμένη έκθεση. Πολλοί συνάδελφοι ήδη είπαν ότι υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση για μια σειρά ζητημάτων που αναφέρονται στην έκθεση. Βεβαίω δεν θα μπορούσαν να συμπεριθούν τα πάντα στο σχέδιο έκθεση, το γνωρίζουμε αυτό. Γι' αυτό έχουμε υποβάλει κάποιε τροπολογίε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία σημεία τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να τονιστούν περισσότερο στην έκθεση. Εμείς θεωρούμε ότι μία από τις αδυναμίες ε, της ΚΕΠΑ το είναι κάτι που αναφέρεται και στον τύπο, αν έτσι το προσλαμβάνει και η κοινή γνώμη, είναι ότι είμαστε πολύ αργοί. Δεν επεμβαίνουμε έγκαιρα. Αυτό έχει να κάνει με τη διαδικασία λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίως θα πρέπει να αλλάξει η συνθήκη. Ε, αλλά και κάποια κράτη-μέλη θα μπορούσαν να είναι πιο προσεκτικά για να έχουμε μια διαδικασία, μια εξωτερική πολιτική που να είναι πιο ευκίνητη. Επίσης πρέπει να γίνει αναφορά κατά τη γνώμη μας στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίζει ρόλο στην θέσπιση της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, Θεωρούμε ότι βεβαίω υπάρχουν κάποια επιτεύγματα τη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία που όμω ε, δεν τα δημοσιοποιούμε επαρκώ, δεν τα διαφημίζουμε. Δηλαδή η κοινή γνώμη δεν ξέρει σχεδόν τίποτα για τα επιτεύγματα τη ΚΕΠΑ. Δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχουν. Καλό θα ήταν λοιπόν κάποια από αυτά να τα γνωστοποιούμε. Επίσης θέλουμε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε, ένα, σε μια διεθνή τάξη που να βασίζεται στο κράτος δικαίου. Και αυτό είναι κάτι που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιπτώσεις ε, κατοχής και προσάρτησης. Παίζουμε διάφορα παιχνίδια ε, και μάλιστα διαφορετικά παιχνίδια ανάλογα με το που βρισκόμαστε ανά τον κόσμο, ενώ πρόκειται για ίδιες καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να να, να αποφασίσουμε αν θέλουμε να έχουμε κάποιες αρχές τις θα τηρούμε πάντα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 15-20 χρόνια οι μονομερείς ενέργειες των Αμερικανών δεν είναι και τόσο εντυπωσιακέ. Όποτε ε, ακολουθούν μια μονομερή ε, πολιτική, τότε η διατλαντική, το διατλαντικό σκέλος της εξωτερικής πολιτικής αποδυναμώνεται και αυτό πάντα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Μέζερης και τώρα για την EFTD ο κύριος Καστάλντο έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ φυσικά για τις προσπάθειες τις οποίες έχετε καταβάλει για την εκπόνηση αυτή της έκθεσης. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, ξεκινώντας από την παράγραφο 5. Έχω κάποιες αμφιβολίες προσωπικά όσον ε, αφορά την ε, αναφορά σε αυτήν την ε, παράγραφο στην ε, μεταναστευτική κρίση και την συμπερίληψη της αναφοράς ότι ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει ένα μίξ αντιμετώπισης ήπιας και λιγότερο ήπιας. Εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τις πραγματικές αιτίες της υποχρεωτικής και αναγκαστικής μετανάστευσης και ενδεχομένως θα πρέπει να βρούμε ένα άλλο ε, ε, σενάριο αν θέλουμε να κάνουμε κάποια αναφορά στο hard power. Στην παραγραφό 8 ε, όσον αφορά τους διαδρόμους και τις, διά, τους διάβλους για την μετανάστευση νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κάποια αναφορά και στις, στην πρόσφατη συνάντηση των τεσσάρων χωρών και ενδεχομένως να πρέπει να γίνει συμπερίληψη και κάποιων άλλων δραστηριοτήτων τον παράγραφος 9. Συμφωνώ απολύτως με παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν κυρίως από τον συνάδελφο Νάρτο όσον αφορά την ε, Ουκρανία και όσον αφορά την αποτυχημένη ε, και λυπή εφαρμογή της ε, συμφωνίας του Μίνσκ. Είναι ιδιαίτερο προβληματική η κατάσταση στη διεθνή σκακέρα και επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να βγούμε από την λογική των κυρώσεων. Θα πρέπει να ξαναρχίσουμε μια προσπάθεια προσπάθεια συζήτησης, διαλόγου με την Ρωσία, γιατί οι αποφάσει αυτέ τελικά γύρισαν μπούμεραν κατά των χωρών μα. Παράγραφος 13 πιστεύω ότι και υπό το φως της παρούσης καταστάσεως ε, σκόπιμο θα ήταν να αναπτυχθεί λίγο περισσότερο το θέμα της ε, απειλής της Βόρειας Κορέας. Ολοκληρώνοντας δε μπορώ να πω ότι για τις παραγράφους 16 και 19 στρατηγική επικοινωνία έχω ισχυρές αμφιβολίες. Νομίζω ότι είναι πολύ ήπιος αυτός ο χαρακτηρισμός που περιγράφει στην ουσία την αντιπροπαγάνδα. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσει τις ανεξάρτητες φορές. Δεν θέλουμε όμως εγγενώς να λέμε το ίδιο και το αντίθετό του. Ο σημερινός κόσμος ε, και χάρη στο ε, ίντερνετ είναι γεγονός ότι έχει φέρει πολλά καλά αλλά έχει δημιουργήσει και το πρόβλημα των fake news, των ψευδών ειδήσεων και επομένως θα πρέπει να είμαστε ε, λίγο πιο προσεκτικοί και θα πρέπει οπωσδήποτε ο λόγος μας να έχει συγκεκριμένες αποχρώσεις έτσι ώστε να μην υπάρξει παρανόηση. Τέλος και πολύ γρήγορα όσον αφορά την, ε, ε, την σημασία του συντονισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 23 και στην, ε, στις κοινέ μάλλον ανταλλαγή πληροφοριών από τις υπηρεσίες πληροφόρησης. Ναι, βεβαίως μπορώ να συμφωνήσω, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει ήδη μεταξύ των κρατών μελών της Ιδίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα πρέπει να αναπτύξουν μεγαλύτερη συνεργασία τα πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα και η αντιτρομοκρατική προσπάθεια συντονισμού μας έχει δείξει το δρόμο. Πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμιστεί περισσότερο η ανάγκη συνεργασίας πρώτα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά ε, με τον ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Φαβίου Καστάλντο. Τσαρλ Στάνοκ ε, από τους ε, συντηρητικού. Ε, ναι, ναι, λέει ο κύριο Τάνοκ. Είχα την δυνατότητα να διαβάσω την εξαιρετική έκθεσή σα Σε παράγραφο 1, επειδή είμαι Άγγλο, πιστεύω ότι αυτό το mentality που γράφεται είναι λίγο υποτιμητικό, έχει λίγο ε, αρνητικό πρόσημα. Ε, θα προτιμούσα κάτι ως perception, αντίληψη, γιατί αυτή η λέξη που έχετε χρησιμοποιήσει είναι υποτιμητική. Δεν συμφωνείτε? Ναι, νομίζω ότι μπορείτε να συμφωνήσετε κι εσείς. Η, η Άννα Γκόμης ε, ε, συμφωνεί στην παράγραφο 8 τώρα. Ναι, καταλαβαίνω την ε, πρόθεσή σας, αλλά εδώ ελοχεύει κίνδυνος να γίνει ένα κορφολόγημα, ένα cherry picking τελικά και ε, τελικά να μείνει η χώρα σε πολύ κακή κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη. Ε, τώρα κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για ε, νόμιμη μετανάστευση αλλά υπάρχει και η παράτυπη και πραγματικά εκεί θα πρέπει να χτυπήσουμε τα αίτια αυτής της μετανάστευσης στις χώρες. Επίσης, ε, είχαμε χθε την συνεδρίαση των ε, πρέσβεων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και είναι περίεργο ε, υπήρξε μια συμφωνία με τη Τεχεράνη, το Ιράν. Ε, πρέπει να ε, γίνει και μια συνάντηση και με την Νότια Κορέα ή Βόρεια Κορέα, συγγνώμη, ή εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική επαφή γιατί έχουμε και τις πρόσφατες βαλιστικές επιθέσεις έναντι της Ιαπωνίας. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης ο Ούγγρος ε, ε, συνάδελφος ε, αναφέρθηκε σε κάποια θετικά στοιχεία της ΚΕΠ. Ας πούμε στην Σομαλία η επιχείρηση Αταλάντη κατά της πειρατείας και να σας πω ότι ήταν επικεφαλής το Royal Navy, το βασιλικό ναυτικό. Εν πάση περιπτώσει ε, ε, κοιτάξτε, ε, υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο και κάνουμε πως δεν τον βλέπουμε και τα πράγματα οπωσδήποτε θα, θα αλλάξουν μετά από το Brexit. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ξαναδούμε συνολικά το θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς ε, ποιος θα είναι ο ρόλος ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ή ποια θα είναι ε, η διαδικασία αναπλήρωσης του ρόλου αυτού. Θα το δούμε μετά. Νομίζω ότι θα πρέπει και εσείς λόγω και της ε, διπλής εθνικότητας να πείτε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει με κάποιο τρόπο στις ε, ε, διαδικασίες. Θα πρέπει έστω και μετά το Brexit επιχειρήσεις τύπου Αταλάντα να συνεχίσουν να λειτουργούν. Υπάρχει μια ολόκληρη στρατηγική, μια ολόκληρη κατασκευή, οικοδόμημα στο οποίο συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν είναι δυνατόν να διαλυθούν όλα με τον Brexit. Ευχαριστώ, Τσάρλ Στάνοκ. Μια σύντομη παρατήρηση. Ε, αρχές Ιουλίου εστάλει η έκθεση και δεν έλαβε υπόψη τις μετέπειτα εξελίξεις στη Βόρειο Κορέα. Όμως θα γίνει αυτό μέσα από τροπολογίες στις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, η ΕΝΕΦ. Ο κύριος Σαφχάουζερ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε αυτή την έκθεση μας λέτε ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε τις εθνικές προοπτικές. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, γιατί οι πολυμερείς ε, ε, σχέσεις θεωρείται ότι έχουν συμβάλει στην ειρήνη. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ρωσία, εάν δεν είχαν αντιταχθεί στην διαδικασία πολέμου στο Ιράκ, ίσως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δεύτερον, μας ζητάτε μια Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίαρχη, αλλά αυτή αποτελείται ε, από κυρίαρχα κράτη. Δεν είναι κυρίαρχη από μόνη της. Ε, κοιτάξτε, εδώ τροποποιείτε τις συνθήκες και εφευρίσκετε νέες ε, συνθήκες. Κάνετε επίσης αναφορά στα ικανότητα, δυνατότητες της Ένωσης. Όχι, είναι οι δυνατότητες και οι ικανότητες των κρατών μελών. Επίσης, λέτε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο χαρακτήρας της ε, ε, ε, αρμοδιότητες και της ουξουσίας. Το σημείο 7 γίνεστε πιο ρεαλίστε. Ε, για την Συρία και τη Λιβύη και σα συγχαίρω γι' αυτό. Αναγνωρίζω ότι η νέα γαλλική πολιτική στον τομέα αυτό είναι πολύ πιο ρεαλιστική και πολύ πιο σωστή ε, και ανταποκρίνεται στην ιστορία και τις παραδόσεις μας ε, και ελπίζω ότι πραγματικά συνέβαλε στη διαδικασία ειρήνευσης στις δύο αυτές χώρες. Επίσης, στο σημείο 9 αναφέρεστε στις κυρώσεις για τη Ρωσία και την κατάσταση στην ε, Ουκρανία. Κοιτάξτε, οι κυρώσει καλό έκαναν μόνο στι Ηνωμένε Πολιτείε. Όσο εμεί μειώνουμε τι ανταλλαγέ μα, μάλλον με την ε, Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε αυξάνουν τι αντίστοιχε συναλλαγέ. Επομένω, νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε αυτό το θέμα των κυρώσεων ε, κατά τη Ρωσία που οι λαοί μα δεν τι θέλουν. Η συμφωνία του Μίσκ, α πούμε, είναι ισορροπημένη. Αλλά τώρα και χάρη στην γαλλική πολιτική και εδώ θέλω να σημειώσω και να υπογραμμίσω τις προτεραιότητες ε, του Προέδρου Μακρόν ε, ε, ανέφερε και αυτός ότι οι, οι συμφωνίες θα πρέπει να είναι ισορροπημένες. Η Ουκρανία έχει μεγάλες ευθύνες για την μη υλοποίηση και εφαρμογή των συνθήκων. Τέλος, εταιρική σχέση με την Αφρική. Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, αλλά εγώ θα ήθελα να επανέλθουμε στις συμφωνίες ΛΟΜΕ, στις συμφωνίες ε, ε, των ε, προτιμησιακών καθεστώτων και όχι στη συμφωνία Κοτονού. Επίσης, ε, αναφέρεστε στον ρόλο της ε, Επιτροπής. Εγώ ε, πρέπει να πω ότι εμείς θέλουμε περισσότερη διακυβερνητική συνεργασία και όχι περισσότερο ρόλο της Κομισιόν και για λόγους καθαρά αποτελεσματικότητας, όχι για λόγους ιδεολειπτικούς. 20-22 έχω ήδη απαντήσει, 23 συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Ναι, εσείς εξισορροπείτε με τις ίδιες δυνάμεις. Πρέπει να πω ότι όντως οι ε, πολίτες μας συμφωνούν με την κοινή άμυνα, αλλά κυρίως ζητούν ανεξάρτητη ευρωπαϊκή άμυνα. Και επομένως θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα της ανεξαρτησίας, γιατί διαφορετικά χάνουμε και την αξιοπιστία μας απέναντι στο ΝΑΤΟ. Επομένως θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω το θέμα της ανεξαρτησίας και των μέσων της Ευρώπης. Άρα, να τα, να, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, άρα τις ικανότητες των κρατών μελών ε, και βεβαίως θα πρέπει να δούμε ε, και το ποσοστό ε, του προϋπολογισμού γιατί το 2% είναι πάρα πολύ λίγο. Επί της εποχής του, Σάρλε, του, του Προέδρου Ντεγκόλ στη Γαλλία είχαμε ποσοστό 4% και επομένως λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες θα έπρεπε να αυξηθεί κατά πολύ το 2%. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Come to Δεύτερος γύρος τώρα αφού μίλησαν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων, έχω πολλούς ομιλητές, 7 συγκεκριμένα, 8 μάλλον. Okay. Um, let's see if we've missed anyone. Θα διαβάσω τα ονόματα. Franca, Mr. Milamon, Mr. Stettin Mr. Preda. From the S&D, Ms. Gomez and Mr. Freund. From ALDE, Mr. Pate. And from the Greens, Mr. Buchner. Διάβασα τα ονόματα από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Και κλείνει ο κατάλογος λοιπόν. Ο κύριος Αλαφράνκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να σας συγχαρώ για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Αντίθετα με αυτά που είπαν κάποιοι συνάδελφοι, εγώ πιστεύω ότι η προσέγγιση για την ασφάλεια είναι απολύτως σωστή και εγγράφεται στις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα η τάση ε, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας είναι μία τάση σαν και αυτή που ακολουθεί η, στρατηγική, η κοινή στρατηγική, όπως λέγει η εκθεσή σας. Δηλαδή, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια, ε, άμυνα, ε, εμπόριο, ασφάλεια, πολιτισμός, όλα αυτά πρέπει να τα συγκεράσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσει που έχουμε μπροστά μας. Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι ότι σε μία έκθεση με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μπορούν να χωρέσουν τα πάντα. Δεν υπάρχει χώρος. Και βεβαίως ε, η έκθεση αυτή μοιράστηκε τον Ιούλιο όπως είπατε, αλλά δεν αποτελούσε μέρος ε, των εγγράφων της Κομισιόν σήμερα, γι' αυτό το διάβασα κάπως, κάπως διαστικά. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια. Ελπίζω να μην έχουν συμπεριληφθεί ήδη στο κείμενο και να μην κάνω λάθος. Αλλά επίσης ήταν πρόεδρος της αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ ε, να αναφερθώ στις προκλήσεις ε, που, δημιουργούνται με τη νέα αυτή κυβέρνηση την Αμερικανική, σε ό,τι αφορά την Ατλαντική Συμμαχία, σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, αλλά και σε άλλου τομεί, όπω το τομέα του προστατευτισμού, η εμπορική πολιτική γενικότερα. Πιστεύω ότι καλό θα είναι να επεκταθούμε εδώ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο βασικό ε, εμπορικό και πολιτικό μα εταίρο. Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε κάπως περισσότερο το ζήτημα αυτό. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην πυρηνική απειλή της Βορείου Κορέας. Είπατε βέβαια ότι όταν συντάχθηκε η έκθεση αυτή δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε τις τελευταίες εξελίξεις ε, με την εκτόψευση πυρηνικών πυράβλων, αλλά θα πρέπει να αναφερθούμε πλέον σε αυτό. Και κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό για μας, διάβασα γρήγορα την έκθεση, αλλά δεν είδα πουθενά καμία αναφορά στη Λατινική Αμερική. Η Λατινική Αμερική, πρόεδρε, είναι ένα σύνολο χωρών που αντιπροσωπεύει το 1 τρίτο των χωρών μελών του ΟΗΕ. Είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά του στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Τρία μέλη της Αμερικής, Λατινικής Αμερικής αποτελούν μέρος του G20. Έχουμε μια έκθεση για την επόμενη συνόδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΑΚ. Ε, υπάρχουν συμφωνίες σύνδεσης με τις οποίες συζητούμε αυτή τη στιγμή ε, Καλό ήταν λοιπόν να γίνει μια αναφορά στα ζητήματα της Λατινικής Αμερικής ε, τα οποία άλλωστε αποτυπώνονται ε, πολύ σωστά στην έκθεση. Ε, κατά τα άλλα η έκθεση σας είναι πολύ καλή. Εμείς θα την υποστηρίξουμε, η πολιτική μας ομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτό το κείμενο που είναι μια καλή βάση για τις εργασίε μας. Όμως έχω και κάποιε παρατηρήσεις, να κάνω κάποιε προτάσεις που ελπίζω ότι θα μπορέσω να τις μετατρέψω και σε τροπολογίες. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να προσποιούμαστε ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Δεν είναι έτσι όσο είναι ο κύριος Τραμπ πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν μπορούμε αυτό να το παρακάμψουμε. Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες. Όχι μόνο για τις σχέσεις μας, αλλά για τον παγκόσμιο ρόλο ε, που θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν οι δυτικέ δυνάμεις ας πούμε και όπως συμφωνούμε με τους Αμερικανούς θεωρητικά θα πρέπει αυτό να το σκεφτούμε ξανά οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε μία έκθεση για αυτό το ζήτημα αγνοώντας ότι υπάρχει αυτή ένας καρκίνος στις διεθνείς σκέψεις στις διεθνείς σχέσεις που είναι η κατοχή της Παλαιστίνης αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε Επίσης ό,τι αφορά τη Λιβύη, συμφωνώ ότι είναι προαπαιτούμενο για την ασφάλεια και στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι στόχος μας, σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση της μετανάστευσης και της αντιμετώπισης τη λαθρεμπορίου ανθρώπων, ε, αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται αναθέτοντας το σε άλλους και να πληρώνουμε εμείς για κέντρα κράτηση στη Λιβύη. Όσο δεν θα υπάρξει πραγματική διακυβέρνηση στη Λιβύη, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν πρόκειται να πετύχουμε αυτό το στόχο. Δεν μπορούμε λοιπόν να ε, στρουθοκαμιλίζουμε. Είναι πολιτικές για τις οποίες ευθύνονται οι δικές μας κυβερνήσεις. Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, Γενικά συμφωνώ, αλλά πρέπει να γίνει και μια αναφορά στη Γεωργία, που επίσης βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες ε, ε, απειλές για την ασφάλεια, την αναφορά στην Αφρική και τη τρομοκρατική απειλή εκεί, καλό είναι να πούμε ότι πολλές από τι προκλήσει έχουν να κάνουν με την έλλειψη δημοκρατικής διακυβέρνησης. Αυτό είναι που οδηγεί στη στρατολόγηση τρομοκρατών ο ρόλος του δίκαιου εμπορίου εδώ είναι πολύ σημαντικός και συχνά τον αγνοούμε. Συμφωνώ επίσης με αυτό που ελέγχθη ότι πρέπει να βρούμε, να πούμε κάτι για τη Βόρεια Κορέα με βάση τις τελευταίες εξελίξεις και απειλές και να πω ότι βεβαίως υπάρχει μια προκλητική στάση, μια επιθετική στάση από την Βόρεια Κορέα αλλά εάν δούμε αυτά που λέει και των ΗΠΑ δεν απέχουν και πολύ σε ό,τι αφορά την αποτροπή τουλάχιστον ενός ε, ε, πυρηνικού ατυχήματος που θα είχε τραγικές ε, επιπτώσεις. Επίσης, την, τις παραγράφους για την ασφάλεια και την άμυνα. Βεβαίως πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τις δυνατότητες της της ασφάλειας και της άμυνας, αλλά είναι σημαντικό λόγω αυτών που είπα για τι ΗΠΑ δεν λέω βέβαια να μην γίνει αναφορά στον ΝΑΤΟ καθόλου αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι σημαντικό να επενδύσουμε στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ανεξαρτησία. Ευχαριστώ την κυρία Γκόμες και τώρα από τους φιλελεύθερους ο κύριος Πάιντε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ε, εγώ την εισηγήτρια και εκπροσωπώ και το σκιώδη εισηγητή μας. Η έκθεση φαίνεται καλή. Είναι θετική η αρχή. Στην παράγραφο 9 γίνεται λόγος για τη Ρωσία ισορροπημένο το κείμενο, το κείμενο, να μην ξεχνάμε ότι είναι επιτιθέμενη η Ρωσία. Συμφωνώ με την Άννα Γκόμες ότι και η Γεωργία θα πρέπει να αναφερθεί εδώ. Παράλληλα, ε, μπορεί να γίνει και επιλεκτική συνεργασία, οπότε αυτό αναφέρεται. Για, ε, επίσης, για την ασφάλεια και τη συνεργασία Ένωσης ΝΑΤΟ, πολύ σωστικά τοποθετείται και υπάρχουν και τα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης που είναι επίσης σημαντικά, αλλά καλό θα ήταν να αναφέρομαι και την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση ε, που προγραμματίζεται σχετικά για το μέλλον. Επίσης, η έκθεση ε, αρχές Ιουλίου δεν αναφέρθηκε όπως έπρεπε στην Βόρειο Κορέα και αυτό θα πρέπει να διορθωθεί, ε, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ευχαριστώ, Τόμας. Ο κύριος Μπούχνερ. Ευχαριστώ πολύ και για την έκθεση αυτή. Ε, καταφέρατε σε 4,5 σελίδες να παρουσιάσετε τα προβλήματα όλου του κόσμου. πραγματικά σας βγάζω το καπέλο. Στο σημείο 8 θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λιβύα, στη Λιβύη, ή αυτό που παρέμεινε από την κυβέρνηση, ε, έχει ε, συνομιλίες σχετικά με το μεταναστευτικό. Οι, εάν επιστραφούν, υποβάλλονται σε βασανιστήρια. Επίσης, ε, ε δημιουργείται μια, ε, ένα, ένας φράχτης ε, βόρεια της Σαχάρας, ε, πράγμα που δεν κατάφερε ο Τραμπ να κάνει και το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κατάφερε να το κάνει ο Τραμπ στο Μεξικό, το κάνει η Ένωση εκεί. Με, με απασχολεί. Αυτό γίνεται και με τα δικά μου ε, χρήματα ε, που δίνω μέσα από τους φόρους. Πιστεύω ότι αυτά ε, τα προβλήματα θα πρέπει να αναφερθούν στην έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Μπούχνερ, ο κύριος Μιλανμόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα γιατί τα είπε και ο κύριος ε, ε, Σαλαφράνκα αυτά που ήθελα να πω. Η έκθεση είναι σωστή, ε, κυρίως όσον αφορά και την εστίαση που κάνει για την τρομοκρατία. Είναι μια πληγή ανοιχτή. Πριν από δύο εβδομάδες μόλις είχαμε το τρομοκρατικό χτύπημα στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Θα πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει έτσι ώστε να καταπληκτήσει πολεμήσει την πληγή του, της τρομοκρατίας και να βελτιώσει και την ζωή των πολιτών. Επομένως, ναι, ε, ε, συμφωνώ με το σημείο αυτό που αναφέρατε. Επίσης, ε, ε, ναι, ε, ε, δίνει το στίγμα μιας αλλαγής, αν όχι νοοτροπίας, αλλά αντίληψης στην, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Επίσης και το γεγονός ότι θα πρέπει οι χώρες να, είναι, να έχουν μια σωστή αντιμετώπιση είναι, συμφωνώ απολύτως και θα πρέπει να δείχνουν την ίδια αξιοπιστία ε, δεν χρειάζεται να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες ε, του κειμένου, ε, γιατί συμφωνώ με τα περισσότερα έτσι αλλιώς. Πιστεύω ότι μια και γίνεται αναφορά στην Αφρική, στην Ασία, θα πρέπει να γίνει αναφορά και στην ε, Λατινική ε, Αμερική. Ε, έχουμε καλές ειδήσει γενικά από τη Λατινική Αμερική, εκτός από το πρόβλημα της Βενεζουέλας. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αναφορά στη Λατινική Αμερική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μιλανμόν. Ο κύριος Φρόιντ. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα σχολιάσω συγκεκριμένα σημεία της έκθεσης. Είμαι ευγνώμων διότι αυτό που ζητούσα από τότε που έγινα ευρωβουλευτής τώρα εκφράζεται σε ένα κείμενο. Ότι δηλαδή χρειαζόμαστε μία ε, αυτοδύναμη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Όπως είπα χθες σε διαφορετική συζήτηση, ως παλιός δημοσιογράφος πάντοτε ενδιαφερόμουν ε, και, ε, ε, για την αναζήτηση της αλήθειας. Και δεν θέλω να παραιτηθώ από την προσπάθειά μου αυτή τώρα που έγινε Ευρωβουλευτής. Άκουσα τον κύριο Σαφχάουζερ να παραπονιέται για τις κυρώσεις ε, που επευλήθησαν στη Ρωσία. Προσθέτω ότι υπήρχε λόγος να γίνει αυτό. Ξεχνάει ότι το 2014 προσήρτησε τη Χερσόν, την ε, Χερσόνησο της Κρυμαίας η Ρωσία και ε, στην Ανατολική Ουκρανία έκανε κρυφό ή μη πόλεμο υπήρχε λόγος για τις κυρώσεις. Μετά ισχυρίζεται ότι οι ΙΠΑ ωφελήθηκαν από τις ευρωπαϊκές ε, κυρώσεις. Εδώ λέω απλώς ότι αυτό δεν αληθεύει. Δείτε τα στοιχεία από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Υπάρχουν στοιχεία. Το 2014 10 δις δολάρια πήγαν στις εξαγωγές και 23 δις στις εισαγωγές από τη Ρωσία. 10 δις προς 23 δις το 2014 λοιπόν. Και τώρα πάμε το 2016, γιατί για φέτος δεν έχουμε στοιχεία. Έχουμε 5 δις και 14 δις αντίστοιχα ε, ε, εξαγωγές εισαγωγές που είναι σχεδόν το μισό. Δηλαδή υποδιπλασιάστηκαν τα στοιχεία ε, εισαγωγών-εξαγωγών σε σχέση με, τη, με τρία χρόνια πριν. Ζητώ λοιπόν από τους συναδέλφους ε, να παρουσιάζουν την αλήθεια πάντα και να μην προσπαθούν να δίνουν εξηγήσεις που δεν έχουν έγκυρη βάση στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ιγκεν Φρόιντ. Ε, ο κύριος Στέτινερ, εμείς θα ακολουθήσουμε τον κατάλογο των ομιλητών σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στα σημεία 9 και 10, καθώ και κάποια άλλα σημεία που έχουν να κάνουν με την Ρωσία. Το σημείο 9 αναφέρεται στη συμφωνία του Μίνσκ. να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία που είχα από την υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ. Συχνά εκεί θέτω το ερώτημα. Υπάρχει κάποιο plan B σε σχέση με τη συμφωνία του Μίντς. Υπάρχει κάποια αναλλακτική σε αυτή τη συμφωνία. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος διαιωνίζεται. Τρία χρόνια έχουν πεθάνει, έχουν σκοτωθεί 10.000 άνθρωποι λόγω αυτού του πολέμου και κανείς δεν ξέρει πώς να το σταματήσει. Εγώ θεωρώ ότι η συμφωνία του Μίνσκ δεν είναι κάποια θαυματουργή λύση και σίγουρα δεν είναι η μόνη λύση. Με βάση την εμπειρία που έχω εγώ από την Ουκρανία. Υπάρχει μια στρατιωτική λύση στο πρόβλημα. Τι εννοώ ο πόλεμος κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να τελειώσει. Και για να τον τελειώσουμε πρέπει να μπλοκάρουμε τα σύνορα των 400 χιλιόμετρων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εάν μπορέσουμε αυτά τα σύνορα να τα κλείσουμε, τότε ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Τι θα γίνει λοιπόν αν αποτύχει η συμφωνία του Μίνσκ. Εντάξει, ακόμα υπάρχει συμφωνία, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να πιέσουμε τους Ρώσους με τις κυρώσεις, όμως η συμφωνία του Μίνσκ είναι τιμοθάνατη όπως και να το κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Ποροσέγκο εδώ και καιρό κάνει εκκλήσεις και στην, στην επέτειο προδημιουργία της Ουκρανίας ε, ζητάει στρατιωτική βοήθεια και έχει δίκιο. Ζητάει βοήθεια για να μπορέσει να κλείσει τα σύνορα με τη Ρωσία. Όταν ο κ. Ποροσέγκο ήρθε εδώ στο Κοινοβούλιο, μα ζήτησε τη βοήθειά μας. Στην έκθεση λοιπόν, θα πρέπει κύριε Πρόεδρε νομίζω, να αναφέρουμε και κάποιες εναλλακτικέ άλλες από, τη Συμφωνία του Μίνσκ που είναι σαφές ότι δεν λειτουργεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Πρεντά, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ζήτησα το λόγο αφού του άκουσα τον κύριο Σαφχάουσερ, ίσως να μιλάει με το λαό στο τηλέφωνο. Ήθελα λοιπόν να σας πω, να πω σε όλους, ότι η ομάδα μου, η πολιτική, υποστηρίζει βεβαίως την θεώρησή σας, την προσέγγισή σας στο έγγραφο αυτό αντίθετα με αυτά που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος από το Εθνικό Μέτωπο της Γαλλίας. Για να βοηθήσω τον κύριο Σαφχάουσερ, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι υπάρχει μια αλλαγή στη ρητορική του, του κύριου Σαφχάουσερ, διότι μέχρι πρόσφατα ο συνάδελφος αμφισβητούσε την Ευρώπη και μάλιστα στο όνομα του λαού έχει αυτήν την, ε, το προνόμιο να είναι ο μόνος που ακούει τη φωνή του λαού. Με αυτό λοιπόν το χάρισμα μιλούσε στο όνομα του λαού, του γαλλικού λαού στην προηγούμενη περίπτωση. Τώρα όμως ε, σταματάει, δεν μιλάει πια για το λαό, μιλάει για τους λαούς. Αναφέρεται στους ευρωπαϊκούς λαούς. Μας λέει λοιπόν ότι υπάρχει κάτι κοινό στους ευρωπαϊκούς λαούς και το, αυτό που ενώνει τους ευρωπαϊκούς λαούς είναι να καταστρέψουν την Ευρώπη. Προ, προηγουμένως το θεωρούσα ότι ίσχυε μόνο για το δικό του λαό, τώρα θεωρεί ότι ισχύει για όλους τους λαούς. Είναι λίγο αντιφατικά όλα αυτά. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε, αυτήν την, σε αυτό το αδιέξοδο και στην αντίφαση για να βοηθήσω τον κύριο Σαφχάουζερ να βάλει κάποια άκρη κάποια στιγμή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, επειδή έγινε φάω ο κύριο Σαφχάουσερ ε, ε, πανελειμμένα ε, προσωπικά έχει το δικαίωμα να απαντήσετε. Ένα λεπτό. Δεν ευχαριστώ περισσότερα, Πρόεδρο. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον φίλο μου, στον τον πω έτσι, τον κύριο Μπρέντα, εμείς δεν είμαστε υπέρ μια, μιας αντιευρωπαϊκής πολιτικής. Εμείς θέλουμε συνεργασία μεταξύ των εθνών και των κρατών. Πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε ότι το εθνικό μέτωπο μεταξύ άλλων είναι αντιευρωπαϊκό. Δεν είμαστε αντιευρωπαίοι. Το έχει πει και η κυρία Λεπέν πολλέ φορέ στην Προεδρική στρατεία. Το είπε. Είμαστε κατά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε κατά τη Ευρώπη. Διότι αυτά τα θεσμικά όργανα δεν λειτουργούν. Αυτά για το πρώτο. Το δεύτερο τώρα. Μου ζητήθηκε να δω τα στοιχεία. Θα σα τα πω. Έψαξα τα στοιχεία σχετικά με τις ε, ε, εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ ε, και Ρωσίας και Ευρώπης και Ρωσίας. Ε, βεβαίως πάντα κανείς μπορεί να ε, παρουσιάζει στοιχεία. Εγώ θα ζητήσω τα στοιχεία τα οποία είχα στη διάθεσή μου στο παρελθόν και θα, θα επανέλθω επ' αυτού. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Άκουσα, προσπάθησα να ακούσω όσο γίνεται πιο προσεκτικά τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ για τα θετικά σχόλια. Θα τα διαβιβάσω στους συμβούλους, που δεν είναι όλοι Πολωνοί, κάποιοι είναι όμως, όπως διαπίστωσε ο συνάδελφος από ό,τι φαίνεται. Ε, ευχαριστώ και για τις ε, πολύ σημαντικές ε, παρατηρήσεις επικριτικές που θα τις ε, λάβω σοβαρά υπόψη και θα βελτιώσουμε την έκθεση μέσα από τροπολογίες. Μία παρατήρηση. Θέλω να υπογραμμίσω άλλη μία φορά ότι παράλληλα ε, τρέχει και μία έκθεση για την ΚΕΠΑΑ που καλύπτει πολλά θέματα ασφάλειας και άμυνας. Για να αποφευθούν οι επικαλύψεις, εγώ προσπάθησα να αποφύγω κάποια θέματα που αφορούν την ΚΕΠΑΑ. Ε, το είπα και στην αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένω τις τροπολογίες σας. Η προθεσμία θα είναι η 12η Σεπτεμβρίου στις 11 το μεσημέρι. Η επόμενη ε, συζήτηση θα είναι 19 Σεπτεμβρίου. 19 ε, Οκτωβρίου, 6 Νοεμβρίου θα γίνει ψηφοφορία και στην Ολομέλεια θα λάβει η χώρα η ψηφοφορία λίγο πριν από τα Χριστούγεννα στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ και πάλι. Και τώρα προχωρούμε στο σημείο 14. Ε, ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να αρχίσουμε τώρα. Ο, ο εισηγητής είναι εδώ. Είναι η ενημέρωση σχετικά με την αποστολή της Επιτροπής ΑΦΕΤ στο Μαρόκο στις, ε, από 17 μέχρι 19 Ιουλίου. Εγώ δεν συμμετείχα στην αντιπροσωπεία. Το καλύτερο είναι να δώσω αμέσως ε, στην αντιπρόεδρο το, στο, ε, στον αντιπρόεδρο το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις εντυπώσεις μας. Ήταν η πρώτη αντιπροσωπεία στο Μαρόκο, παρόλο που είχαμε συναντηθεί με τους Μαροκινούς σε άλλες περιπτώσεις, σε, ε, στο παρελθόν. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν στο ταξίδι. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η αντιπροσωπεία και όλοι συνέβαλαν εξαιρετικά στις συναντήσεις με τους Μαροκινούς. Ευχαριστούμε και τους εκπροσώπους από την ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων για τη συμμετοχή. Γενικά πρέπει να πω ότι οι συναντήσεις της αντιπροσωπείας μας ήταν υψηλού επίπεδου, ήταν τον Πρωθυπουργό, τον ΙΠΕΞ, τον υπεύθυνο Υπουργό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Ήφη Υπουργό Δικαιοσύνη και άλλου ε, είδαμε τον ένα πρόεδρο του ενός κοινοβουλευτικού σώματος δηλαδή, έχει δύο σώματα. Ε, επίσης δώσαμε την πρόσκληση στον ΙΠΕΞ από τον πρόεδρο να έρθει το φθινόπωρο σε, στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και να ανταλλάξει ε, απόψεις με την Επιτροπή. Ο απεδέχθη την πρόσκληση και τώρα ε, ρυθμίζονται ε, τα πρακτικά θέματα με τις υπηρεσίες. Ένα ε, θέμα που είδαμε είναι ότι υπάρχει μια μετατόπιση στην εκπροσώπηση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης στο Μαρόκο. Ο επικεφαλής και ο αναπληρωτής του έφευγαν ε, θα για να αντικατασταθούν. Αυτό ήταν λίγο ατυχές, γιατί άμα ήταν εκεί θα είχαμε ενημερωθεί πολύ καλύτερα, θα μπορούσε να είναι δηλαδή και ο ε, απερχόμενος και ο επόμενος. Δεν έγινε όμως αυτό. Εμείς ε, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πάντως ε, υπήρχε εκπροσώπηση από την αντιπροσωπεία σε όλο το ταξίδι. Κάποια θέματα τώρα που μας απασχόλησαν με τους Μαροκινούς. Το Μαρόκο ξέρετε ότι είναι από τις χώρες με τις οποίες έχουμε ε, πολλά θέματα που συζητήσει σε βάθος, συνεκτικά. Οι συναντήσεις μας καλύπτουν πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι το εμπόριο. Επίσης ε, μιλήσαμε με το, για το θέμα της ε, ε, Δυτικής Σαχάρας και το, την απόφαση του δικαστηρίου. Επίσης ε, είδαμε τον επικεφαλής των ανεξάρτητων, της, της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και παρουσιάσαμε και ορισμένε απόψεις της Ένωσης. Η μετανάστευση, η καταπολέμηση τρομοκρατίας σε μεγάλο βαθμό καλύφθηκαν επίσης Συνολικά λοιπόν μπορώ να πω ότι είχαμε ένα ευρύ φάσμα συζητήσεων επί όλων των ε, θεμάτων και στα διαφορετικά επίπεδα. Και είχαμε και πολύ εκτενή κάλυψη της επίσκεψής μας από τα ΜΜΕ. Συνολικά πρέπει να πω ότι η ε, αποστολή πέτυχε το στόχο της να ε, συνεννοηθεί με τους Μαροκινούς σε κυβερνητικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο και καλό είναι να ε, δώσουμε συνέχεια όταν συναντήσουμε τον υπέξ τον Μαροκινό στην Επιτροπή ε, αυτή αργότερα μέσα στο χρόνο. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την καλή τους συνεισφορά και το πνεύμα συνεργασίας τους που σημαίνει ότι μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς το βαρύ πρόγραμμα. Τέλος, ε, περάσαμε μία μέρα και στην Καζαμπλάνκα, όπου καλύψαμε κάποια θέματα εμπορικά με τα διάφορα εμπορικά επιμελητήρια από τις διάφορες χώρες και ε, ε, κάναμε και ένα ταξίδι όπου επισκεφθήκαμε επιτόπου κάποιους ε, φορείς ε, που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο. Και ήταν πολύ θετικό αυτό και ήταν μια ωραία κατάληξη της επίσκεψης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιστήσεν. Ε, επιβεβαιώνω ότι έχει αποσταλεί πρόσκληση προς τον Πρωθυπουργό του Μαρόκου ε, για τον ε, Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε τώρα τις παρεμβάσεις με την ε, κυρία Γιάλα Σέντερ, η οποία είναι αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας με το Μαρόκο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ε, η οποία έδωσε την ε, δυνατότητα ε, να συμμετάσχει η πρόεδρος αντιπροσωπείας για τις χώρες Μαχρέμπ σε αυτήν την ε, αποστολή. Είναι πολύ καλός αυτός ο τύπος συνεργασίας ε, μεταξύ, στις αποστολές ε, μεταξύ επιτροπών και αντιπροσωπιών. Εγώ προσυπογράφω τόσο είπε ο κ. Βίστησαν όσον αφορά την καλή ε, ε, εξέλιξη των εργασιών της ε, αποστολής που ήταν μάλιστα και υψηλού επίπεδου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω κάποια σοβαρά θέματα και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό που ο Υπουργό αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόσκλησή μας και θα είναι σίγουρα πολύ θετική η ανταλλαγή απόψεων. Θα είναι καλό να είμαστε παρόντες. Επίσης σημαντικό σημαντική νομίζω ήταν ε, η παρουσίαση που μας έγινε ε, της, ε, του νέου δικαστικού συστήματος του Μαρόκου που είναι η πραγματικά μεγάλη μεταρρύθμιση που λαμβάνει τώρα χώρα και στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας Επίσης συζητήσαμε ε, σε μια πολύ σημαντική ε, στιγμή που μας απασχολούσε ε, ιδιαίτερα το θέμα των αντιδράσεων ε, και ε, η προβληματική ε, κατάσταση η οποία προκύπτει από τις μεγάλες διαφορές, περιφερειακές διαφορές. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε και με τους υπουργούς και μετά από την απόφαση του δικαστηρίου. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε σημείο και σε σημαντική στιγμή οι σχέσεις με το Μαρόκο. Ε, είχαμε την αίσθηση ότι προχωρούν τα πράγματα προς την καλή, ε, προς μια σωστή κατεύθυνση. Επίσης, όταν θα έρθει ε, ο υπουργό Εξωτερικών, καλό θα είναι να τον ρωτήσουμε για τον ρόλο που προσπαθεί να αναπτύξει το Μαρόκο σε σχέση με την κρίση της Λιβύης. Τέλος ένα αρνητικό στοιχείο, όχι ακριβώς αρνητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει αρνητικό πρόσημο ας πούμε. Η ορατότητα ε, της ε, συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ε, σημαντική γιατί γίνεται μέσα από συγκεκριμένη γραμμή του περιπολογισμού. Αυτή η συνεργασία δεν φαίνεται πάρα πολύ. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να αυξηθεί η ορατότητα. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αγιάλα Σέντερ. Βλέπω μια ανακοίνωση εδώ, μόλις πληροφορηθήκαμε ότι, ότι δεν έχουν λάβει επίσημη πιστοποίηση οι ε, ε, πρέσβεις μας ε, στην Βενεζουέλα στο Μαρόκο δεν θα, έχουν τη δυνατότητα να είναι μαζί μας αύριο για την ανταλλαγή των απόψεων. έχουμε, θα έχουμε όμως πάντα μαζί μας τον νέο πρέσβη στην Μόσχα. Οπότε εντάξει τουλάχιστον για αυτόν. Ο κύριος Πρέντα και αυτός ήταν στην ομάδα της αποστολής. Ευχαριστώ πολύ. Um, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Μαροκινούς, ε, την Μαροκινή πλευρά για την υποδοχή που μας επεφύλαξαν. Και μάλιστα αφού φέτος είχαμε κάποιες εμπειρίες λίγο οριακές με την υποδοχή που μας επεφύλασαν ε, ε, οι αντίστοιχες πλευρές σε κάποιες αποστολές μας εδώ. Είχαμε όμως μια πολύ καλή επαφή, είχαμε πολύ ε, καλούς και υψηλού επίπεδου συνομιλητές, υπουργούς, ε, και ανθρώπους που είδαμε ότι πραγματικά είχαν ενδιαφέρον ε, να συζητήσει μαζί μας. Ας πούμε, ε, μια μισή ώρα κράτησε η ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Δικαιοσύνης ε, μία, ε, και μάλιστα μας είπαν ότι ε, η πρώτη φορά, πρώτη φορά είχαν μία αποστολή από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Είχαν βεβαίως αποστολές και επισκέψεις της αντιπροσωπείας για το χώρες Μαχρέμ και τα λοιπά, αλλά εδώ από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πρώτη φορά. Άκουσα προσεκτικά λοιπόν του συνομιλητές μας και έχω εξάγει κάποια συμπεράσματα. Πρώτο συμπέρασμα συνδέεται με το θέμα της μετανάστευσης, διότι στις ανταλλαγές που είχαμε ε, με τους πολιτικούς συνομιλητές μας, σε μια εξαιρετική συνεδρίαση που είχαμε με τους εκπροσώπους ε, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Ε, καταλάβαμε πάρα πολύ καλά ορισμένα πράγματα. Ε, το Μαρόκο δεν είναι χώρα από την οποία ξεκινά μετανάστευση. Δεν είναι χώρα διέλευσης μεταναστών, είναι πλέον χώρα στόχος, χώρα υποδοχής. Και δεν είναι και η μόνη χώρα. Ας δούμε τι γίνεται στην Αλγερία, τι γίνεται στην Τινησία. Αυτές οι χώρες ε, Μαγρέπ διαπιστώνουν σήμερα ότι πλέον έχουν γίνει ε, ε, πραγματικοί στόχοι μετανάστευσης. Η χάρια μετανάστευση σταματά στις χώρες αυτές και επομένως θα πρέπει λίγο να ξαναδούμε τις, τις πολιτικές που εφαρμόζουμε εκεί και τις δράσεις μας. Δεύτερο συμπέρασμα σχετικά με τον πολιτικό Ισλαμισμό είναι ένα ζήτημα το οποίο πολύ μας απασχόλησε μετά από την Αραβική Άνοιξη. Αλλαγέ, ε, αρχίσαμε να ρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε με τον πολιτικό Ισλαμισμό. Πρέπει να πούμε στο Μαρόκο, η κύρια, ε, το, το κύριο ε, κυβερνητικό άλλωστε κόμμα ορίζει, λέει ότι είναι Ισλαμικό. Στην ουσία, αυτό που, ε, η προσπάθεια που κάνει το Μαρόκο είναι να φημώσει κατά κάποιο τρόπο τον Ισλαμισμό ε, έτσι ώστε ε, το κόμμα PZD να συμμετάσχει στην κυβέρνηση μαζί με άλλες πολιτικές ομάδες. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία μία κυβέρνηση συμμαχίας που αποτελείται από 7 διαφορετικά ε, κόμματα. Και επίσης να πούμε ότι κάποιες πολιτικές όπως ας πούμε ε, η πολιτική για τις γυναίκες δεν είναι πάρα πολύ εύκολη ε, και δεν είναι δυνατό να συμφωνηθεί εύκολα όταν ας πούμε ο αρμόδιος υπουργός είναι Ισλαμιστής. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε χαόδη κατάσταση στο Μαρόκο όπως βλέπουμε σε άλλες ε, χώρες ε, στη Λιβύη και σε άλλες χώρες της ε, περιοχής που ορίζουν την πολιτική τους θέση ως θέση καθαρού Ισλαμισμού. Εδώ στο Μαρόκο είδαμε ότι έχουμε πολιτικά κόμματα με παραδοσιακούς πολιτικούς ιδεολογικούς προβληματισμούς. Τρίτον, είχαμε εξαίρετη συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος μας ανέφερε ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για τις ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή την επιστροφή των Ισλαμιστών που έχουν πάει στην Συρία ή στο Ιράκ ε, για να αγωνιστούν για το Χαλιφάτο στο Μαρόκο λοιπόν προς ώρας έχουν καταγράψει περίπου 1.600 επιστροφές στο Μαρόκο, επί των οποίων 400, 400 είναι παιδιά. Ε, δηλαδή το 1 τέταρτο των επιστροφών ε, είναι παιδιά. Αυτή την καταγραφή έχουν κάνει οι μαροκινές αρχές. Μας έδωσαν και κάποιες ε, ε, λεπτομέρειες ε, γιατί πραγματικά ασκούν μια πολιτική απορριζοσπαστικοποίησης και έχουν και μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση των στρατιωτών ας πούμε, του Χαλιφάτου που επιστρέφουν. Αυτά είχα να πω και σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλή συνεργασία με συναδέλφους άλλων ομάδων. Thank you. Christian Ευχαριστώ τον Κρίστιαν Πρέντα και τώρα και ο Σπαντζέρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν θέλω να προσθέσω και πολλά γιατί όλα έχουν υποθεί. Απλώς θα ήθελα να επαναλάβω ένα πολιτικό στοιχείο. Είναι απολύτως προφανές ότι το Μαρόκο στα πλαίσια της Βόρειας Αφρικής είναι μία χώρα που μπορούμε να πούμε ότι είναι μάλλον φυσιολογική σε αντιπαράθεση με δύσκολες ε, καταστάσεις σε άλλες χώρες όπως η Λιβύη, ε, δύσκολη μετάβαση στην Τινησία, προβλήματα στην Αλγερία τα οποία ε, είναι κρυμμένα αλλά υπάρχουν. Επομένως είναι γεγονός ότι μπορούμε να, ότι πρέπει να κάνουμε μια σωστή δίκαιη αξιολόγηση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα αυτή, αυτό το διάστημα. Ε, είναι απαραίτητο ε, να συνεχίσει ε, η διαδικασία πολιτικής μεταρρύθμισης. Το θέμα της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης που είναι ευαίσθητο θέμα ή το θέμα των περιφερειών που έχει ξεκινήσει να αντιμετωπίζεται αλλά εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Το θέμα της περιφερειοποίησης το οποίο ο Σένφος πρέπει να έχει παρακολουθήσει είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και το οποίο συνδέεται και με την, ε, ε, την ε, Δυτική Σαχάρα και επομένως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει ειρήνευση στην περιοχή. Κοιτάξτε, εμείς δεν είδαμε ε, ε, εμείς δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Όντως, ε, στην περιοχή της Ταγκέρης έχουμε ζυμώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Στο Βόρειο Μαρόκο έχουμε έτσι έναν αναβρασμό και αυτό που είναι γεγονός είναι ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή έτσι ώστε αφενός να την βοηθήσουμε στη διαδικασία μεταρρύθμισης αλλά και από την άλλη πλευρά να ε, μπορέσουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε οι προσδοκίες του μαροκινού λαού να μην διαψευστούν. Ε, θα πρέπει και εδώ να πούμε ότι ε, είναι ιδιαίτερα συντηρητική η διοικούσα τάξη του Μαρόκου. Του Μαρόκου. Είναι τύχη και το βάζω εντό εισαγωγικών ότι ο Μοχάμετο έκτος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την ε, διοικούσα και την άρχουσα τάξη και επομένως ε, ε, υπήρξε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί καλύτερα, να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι προσδοκίες του λαού του Μαρόκου. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε όμως, θα πρέπει να προσέχουμε έτσι ώστε να δοθεί η απαραίτητη όθηση για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία μεταρρύθμισης. Ευχαριστώ κυρία Λαλόντα από τους φιλελεύθερους. Έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με όλα όσα ελέγχθησαν. Η αποστολή αυτή ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πολύ καλά οργανωμένη. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Πέντρα Ήθελα απλώς σε σχέση με την ε, ε Ισλαμοποίηση και τον εξισλαμισμό να πω κάτι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο στο Μαρόκο ε, να διαχειριστεί κανείς την κατάσταση. Εγώ πάω εδώ και χρόνια στο Μαρόκο ε, και υπάρχει Ισλαμοποίηση. Η διαφορά είναι τεράστια σχέση με πριν από 15 χρόνια. Αυτό μου το είπαν και ΜΚΟ, για τα δικαιώματα των γυναικών, οι γυναίκες μου εξηγούν ότι, τα, ότι υπάρχει τεράστια πιστοδρόμηση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους. Συναντήσαμε βεβαίως τον Υπουργό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αποτελεί μέρος του PGD που προσωπεί το πολιτικό Ισλάμ και που είναι βεβαίως όμως ταυτόχρονα κοντά ε, στους αδερφούς μουσουλμάνους. Ήταν πολύ συμπαθητικός, ε, του εξηγήσαμε μια σειρά πράγματα, όμω του ρωτήσαμε για τους πρόρους γάμους στο Μαρόκο μας είπε βεβαίως ότι θα υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, ότι είναι κατά, αλλά μας εξήγησε ότι ξέρετε υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και βέβαια ο διάβολος κρύβεται πάρα στις λεπτομέρειες και στις εξαιρέσεις αυτές μας είπε ότι πιο φτωχοί σε κάποιες περιοχές της χώρας έχουν την τάση να ε, θελήσουν να παντρέψουν τη μικρή τους κόρη, ε, μας από από λεπτομέρειες τώρα, αλλά είναι αρκετά σοβαρό θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου το γνωρίζει αυτό, κάνει ό,τι μπορεί, αλλά είναι σημαντικό, εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση, αυτή η οπισθοδρόμηση, αυτή, αυτός ο εξισλαμισμός ε, της ε, κοινωνίας είναι πολύ περισσότερες οι γυναίκες ε, που φορούν ε, μαντήλα στις μεγάλες πόλεις, στη Ραμπάτ, στην Καζαμπλάνκα και βεβαίω υπάρχει το θέμα τη τρομοκρατία. Ε, είχαμε και τη Βαρκελόνη. Έκτοτε με μια μαροκινή ε, έτσι, ομάδα τρομοκρατών. Ξέρουμε ότι το Μαρόκο κάνει τεράστια προσπάθεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί, είναι και υποδοχή, χώρα υποδοχή μεταναστών από την υποσχάρια Αφρική, αλλά πρέπει να επαγρυπνούμε. Όπω είπε και ο κύριο Πέδρα, είναι όλοι αυτοί οι μαχητέ από το Ιράκ και τη Συρία που επιστρέφουν. Ε, στο Μαρόκο αυτή τη στιγμή. Το γνωρίζει αυτό η κυβέρνηση βέβαια. Καλό, ήταν, καλό είναι πάντως να γίνει ένα φόρο στα δικαιώματα των γυναικών διότι είναι πραγματικά σοβαρή η κατάσταση. Δεν αφορά βέβαια μόνο το Μαρόκο αυτό, αλλά και το Μαρόκο. Um, um, Ευχαριστώ. Έχουμε πέντε ομιλητές ακόμα. Mr. Sole and Mr. Buchner. Did we miss somebody? Ε, τους ανέφερα όλους, ναι. Οπότε τρία λεπτά θα δώσω στον καθένα. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Σόλε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήταν πράγματι ενδιαφέρουσα αποστολή. Με πολύ βαρύ πρόγραμμα. Όμως, συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ήδη. Ήθελα μόνο να ε, τονίσω κάποια πράγματα. Πήγαμε στο Μαρόκο σε μια σημαντική στιγμή για τη χώρα αυτή, όπου η κρίση ε, εξελίσσεται στο βόη. Ε, παίζει ρόλο στη, στο χώρο Μαγκρέμπ και στη νότια γειτονία της Ένωσης και είναι και μια χώρα που παλεύει για να ε, εφαρμόσει πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα εδραιώσουν το δρόμο προς τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Συγκεκριμένα θέλω να παρουσιάσω μια εντύπωση, μια αίσθηση που αποκόμισα μετά από πολλές συναντήσεις με υπουργού και σίγουρα και με τον Πρωθυπουργό, γιατί ε, πήγαμε σε σημαντική στιγμή στο Μαρόκο και για τις σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Μαρόκου, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του περασμένου Δεκεμβρίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών στη Δυτική Σαχάρα και σε πολλές συναντήσεις μας ε, ε διαισθάνθηκα ότι υπήρχε κάποια απογοήτευση ε, των μελών της κυβέρνησης σχετικά με το πώς προσεγγίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το Μαρόκο. Όταν ρώτησα τον Πρωθυπουργό, για παράδειγμα, τι πιστεύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι ε, δέχεται και αναγνωρίζει ότι είναι βασικός ε, φίλος του Μαρόκου η Ένωση, αλλά θέλει ε, να κάνει περισσότερα η Ένωση για να αναγνωρίσει τις προσπάθειες του Μαρόκου, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Επίσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης παραδέχτηκε ότι υπάρχει μια απογοήτευση στην κοινή γνώμη σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει η Ένωση το Μαρόκο. Το Μαρόκο γνωρίζει καλά τη σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι πύλη προς την Ευρώπη, είναι σημαντικός οικονομικός εταίρος και είναι και εταίρος στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Παράλληλα όμως ε, θεωρούν ότι υπάρχει μια έλλειψη ενδιαφέροντος από ευρωπαϊκής πλευράς και αυτό έχει σχέση και με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ελπίζω να βρεθεί μια καλή λύση σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση του Δικαστηρίου. Αλλά θα πρέπει να, να ακουστούν και οι δύο πλευρές. Ε, πρέπει να ε, λυθεί το θέμα της Δυτικής Σαχάρας και ε, να κατησχύσει η αρχή της αυτοδιάθεσης. Όλα αυτά πρέπει να τύχουν επεξεργασίας για να βελτιώσουμε τη σχέση μας με το σημαντικό εταίρο Μαρόκο και τελειώνω λέγοντας ότι ε, δεν είναι θετικό ότι δεν έχει διαπιστευθεί ο, ε, η αντιπροσωπεία μας στο Μαρόκο. Δεν είναι καλό δείγμα αυτό. Και θεωρώ ότι δεν βοηθάει την όλη κατάσταση. Ευχαριστούμε. Τον Πράφκα Σουίτσα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ε, των επικεφαλής αντιπροσωπείας που ήταν πολύ καλή αντιπροσωπεία και με τον κύριο Παντσέρη και με αντιπρόσωπο, εκπρόσωπο από την Επιτροπή Γυναικών. Ο στόχος ήταν να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο και παράλληλα όπως ακούσατε είχαμε σοβαρές και υψηλού επίπεδου συναντήσεις. Εγώ θέλω να τονίσω το, τη ριζοσπαστικοποίηση και την καταπολέμησή της που είναι πολύ σημαντικό, η μετανάστευση, θέματα φύλου, πολύ σημαντικά, ισότητας. Δεν είδαμε γυναίκα σε υψηλά αξιώματα, ούτε μία, μόνο σε διοικητικές θέσεις ήταν γυναίκες. Δεν ε, είδαμε ε, σε ηγετικέ θέσει γυναίκες. Αυτό είναι προβληματικό. Και αυτό που συμπεραίνω από τη συνάντηση αυτή είναι ότι η προκήρυξη μεταρρυθμίσεων είναι ένα πράγμα και η εφαρμογή τους άλλο. Ε, χρειάζονται βοήθεια εδώ, προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν και το σημαντικό είναι η Δυτική Σαχάρα και η απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να εφαρμόσουν την απόφαση, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Δεν προβλέπω ότι θα είναι εύκολη η εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Περιμένω να έρθει ο υπέξ εδώ στην Επιτροπή μας για να συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ, Ντουμπράφκα. Ο κύριος Παρνιό. Κύριε Πρόεδρε, να πω και εγώ δύο λόγια εν συντομία. Πρώτα απ' όλα, όντως συναντήσαμε τις πολιτικές αρχές του Μαρόκου σε υψηλό επίπεδο και αυτό είναι σημαντικό στα πλαίσια αυτής της πρώτης επίσκεψης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερον, εδώ και κάποια χρόνια συμμετέχω σε αυτές τις συναντήσεις ε, εταιρική σχέση με τους μαροκινούς φίλους και πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθω εκ μέρους των μαροκινών αρχών ομόφωνα, ε, ομόθυμα μια κάποια απογοήτευση. Έχουν την εντύπωση ότι δεν αναγνωρίζεται η θέση τους από την Ευρώπη. Δεν την χάνουν αναγνώρισης. Όχι μόνο από εμάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ιδίως ό,τι αφορά τρεις πολιτικές. Πρώτα, το θέμα της μετανάστευσης. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Πρέντα. Το Μαρόκο έχει μετατραπεί σε χώρα προορισμού και έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές ροές τις τελευταία χρόνια, τις τελευταίους μήνες μεταναστευτικές ροές από την υποσοχάρη Αφρική, οι οποίες δεν δείχνουν να μειώνονται. Θα πρέπει λοιπόν εμείς ως Ευρώπη να το εξετάσουμε αυτό το ζήτημα προσεκτικά, για να μην υπάρξει αποσταθεροποίηση σε μια πολύ σημαντική χώρα όπως το Μαρόκο, ε, εντός αυτού του πολιτικού και οικονομικού πλαισίου ε, στο Μαγκρέμπ και στην Αφρική. Δεν πρέπει να προσταθεροποιηθεί το Μαρόκο. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν πολύ προσεκτικά την εταιρική μας σχέση σε σχέση με τα μεταναστευτικά ζητήματα. Δεύτερον, θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης πολύ προσεκτικά το θέμα της πρόληψης ε, της ριζοσπαστικοποίησης. Η θέση της, ε, του, της θρησκείας γενικότερα στην κοινωνία ε, και στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Το μετριοπαθές Ισλάμ είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε για να αποφύγουμε ακριβώς αυτό το πολιτικό Ισλάμ, για να αποφύγουμε τον εξισλαμισμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών, όπως είδαμε με τις ακρότητες τις οποίες διαπιστώνουμε και που δυστυχώς ε, διαπιστώσαμε εκ νέου αυτό το καλοκαίρι στη Βαρκελόνη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό εδώ, στα πλαίσια της καταπολέμησης τρομοκρατίας, απέναντι στη ζωσπαστικοποίηση, να συνεχίσουμε εμείς να αναπτύσσουμε την εταιρική μας σχέση με το Μαρόκο. Και τέλος, θα πρέπει να αναπτυχθεί η εταιρική μας σχέση και η συνεργασία μας για ζητήματα οικονομικά και κοινωνικά, ζητήματα αν μια ελλειπούς οικονομικής ανάπτυξης στο Μαρόκο, ε, μια ε, ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, την κοινωνική προστασία, η μείωση των ανισοτήτων. Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και εδώ θα πρέπει να απαντήσουμε στις προσδοκίες του Μαρόκου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Παρνιό και τώρα θα δώσω το λόγο σε δύο συναντρέφους που δεν ήταν στην αποστολή αλλά που θέλουν να παρέμβουν. Πρώτα ο κύριος Νάρτ και μετά ο κύριος Μπούχνερ. Κύριε Νάρτ, έχετε το λόγο. Το Μαρόκο είναι σίγουρα η καλύτερη χώρα της Βορείου Αλλά έχει και τεράστια προβλήματα όταν λέμε ότι επισκεπτόμεθα τους πολιτικούς του Μαρόκου, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής του Μαρόκου ελέγχεται από το παλάτι, από το βασιλιά, διότι υπάρχουν υπουργεία τα οποία είναι δική ορμοδιότητα, τα πιο σημαντικά, άμυνα, ασφάλεια, εξωτερική πολιτική κτλ. Ε, δηλαδή δεν είναι απλά ο βασιλιάς του Μαρόκου, είναι και επικεφαλής ε, των πιστών, έχει ένα θεακροατικό χαρακτήρα. Επίσης, το μεγα... η, η δυναστεία των Αλαουίτων είναι αυτή που έχει τα περισσότερα χρήματα, τις μεγαλύτερες περιουσίες. Δεν είναι μόνο θέμα λοιπόν κάποιων μεταρρυθμίσεων. Διότι εδώ μιλάμε για κάποιες καλλιτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ υπάρχουν κάποια τεράστια προβλήματα. Μία νεολαία που είναι εκτός συστήματος, πρώτον, και δεύτερον, μία κατάσταση Ισλαμισμού που κάποιοι ονομάζουν ε, μετριοπαθές, αλλά υπάρχει ε, ε, και μια άλλη τάση που, που ονομάζεται δικαιοσύνη και θρησκεία. Ε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι λοιπόν ε, τρομοκράτες στην Ευρώπη είναι μαροκινής προέλευσης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη παρουσία μαροκινών τζιχαντιστών και στο Ιράκ και στη Συρία. Δηλαδή, αναλογικά με άλλες χώρες, είναι μεγάλα τα ποσοστά. Πρέπει να τα λέμε όλα. Επαναλαμβάνω, είναι η καλύτερη χώρα της Βορείου Είναι μια κρίσιμη σημασία χώρα για μας, για ζητήματα που έχουν να κάνουν στην περιφερειακή σταθερότητα, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη μετανάστευση. Αλλά, και πρέπει να το πούμε αυτό, και είναι θετικό, αλλά προσοχή. Δεν πρέπει απλά να μένουμε θεατές προ κάποιων καλλιντικών μεταρρυθμίσεων επουσιοδών, ενώ έχουμε μια πολιτική σχιζοφρένεια, όπου η πραγματική εξουσία, η ουσιαστική και η οικονομική βρίσκονται στα ίδια χέρια. Ε, χαίρομαι που υπάρχει ρεαλισμό από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, από τη Γαλλία, από την Ισπανία, στη σχέση με το Μαρόκο. Η κατανόηση απέναντι στο θέμα τη Δυτική Σαχάρας όπου κάνουμε κάποιες δηλώσεις μεταφυσικές εντελώς. Ε, είναι πραγματικά ευχολόγιο, τίποτα άλλο. Για να μην πούμε στην ουσία του ζητήματος. Διότι η ουσία του ζητήματος ε, ίσως να είναι και χειρότερη για την Ευρώπη από ό,τι για το Μαρόκο. Πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Πέρα από αυτά που δηλώνουμε επισήμως. Επιμένω, αυτός ο ρεαλισμός είναι σημαντική, σημαντικός ε, απέναντι σε μια χώρα τόσο σημαντική για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ισπανία. Θα πρέπει λοιπόν αυτός ο ρεαλισμός ε, να πρεσβεύει και αλλού, όπως παραδείγματος χάρη στη σχέση μας με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούχνερ τέλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εκπλήσωμαι που σε όλες αυτές ε, τις εκθέσεις, οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα δεν αναφέρθηκαν γιατί γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό του Μαρόκου, αλλά στη Δυτική Σαχάρα είναι πολλές οι ομότητες. Ε, ως Ευρώπη δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ε, ανοιχτά ότι την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα την παρακάμψει όσο γίνεται επειδή οι business είναι πολλές και καλές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο, να δώσουμε περισσότερη έμφαση στις αρχές μας εν προκειμένου. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ ευχαριστώ συνάδελφοι για την συμβολή σας. Δεν βλέπω να ζητεί άλλο το λόγο. Οπότε προχωρούμε στο σημείο 15 και καλωσορίζω τον κύριο Αλεξάνδερ Ρόντος. Ελάτε ε, εδώ μπροστά παρακαλώ. sundowner and smoking. so, thank you. λοιπόν, αγαπητοί μου συνάδελφοι, είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να καλωσορίσω τον κύριο Αλέξανδρο Ρόντο. Καλησπέρα. Συνήντησα πριν από τέσσερι εβδομάδε τον Αλέξανδρο Ρόντο στην αποστολή παρακολούθηση των εκλογών στην Κένια. Είναι ειδικό εκπρόσωπο στο κέρας της Αφρικής. Ο κύριος Ρόντος ήδη είναι έξι χρόνια στη θέση αυτή. Είμαστε πολύ ευτυχείς που θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων σήμερα στο φως της εκτενούς αυτή την περιοχή με τις πολλές προκλήσεις. Καλύπτει τη Σομαλία, το Σουδάν, Νότιο Σουδάν, Τζιμπούτι, Ουγκάντα, Ερυθρέα, Αιθιοπία, Κένια, Σομαλία, Τζιμπούτι. Ήταν καλή ιδέα να ε, προσκαλέσω με τον κύριο Ρόντο εδώ γιατί μας μίλησε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές σε μια εκδήλωση για πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε την περιοχή, ε, στη Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Σουδάν. Ε, ο πόλεμος ε, έχει μεγάλο τίμημα, αποσταθεροποιεί όλη την περιοχή. Για χρόνια υπήρχαν μεγάλα προβλήματα και μετανάστευση από την Ουγκάντα. Υπάρχουν και θέματα συνόρων μεταξύ Αιθιοπίας, Ερυθρέας, Σουδάν, Νότιο Σουδάν. Η Εμένη επίσης τώρα... Ε, και η στάση της στο μεταναστευτικό μπορεί να δημιουργήσει θρησκευτικέ εξάρσεις πάλι. Ε, Πολλές είναι οι εξελίξεις λοιπόν στο κέρας Αφρικής. Χαίρομαι που θα μας ε, ενημερώσετε. Ελπίζω να μας πείτε εκτός από τις προκλήσεις και κάποιες θετικές εξελίξεις που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Και είμαι πεπισμένος ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσέχουμε και να, στο μέλλον ακόμη περισσότερο να προσέξουμε αυτή την περιοχή του κόσμου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ David. Ήταν μεγάλη μου χαρά που σε είδα στο Ναϊρόμπι με κάποιου συναδέλφους Φουσουσού λίγο πριν από τις εκλογές. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για να ανταλλάξω απόψεις με όλους εσάς. Όπως είπα στον Ντέιβιτ και τους συναδέλφους τους, τους άλλους ευρωβουλευτές, είμαι ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει όλης της Ένωσης που περιλαμβάνει και αυτό το Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν πάντοτε χαίρομαι να βρίσκομαι στη διάθεσή σας. Για λόγους χρόνου, εξοικονόμησης χρόνου, θα είμαι πολύ ε, σύντομος εγώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις που είμαι βέβαιος ή τουλάχιστον ελπίζω να έχετε. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις πρώτα για την περιοχή αυτή. Ε, γνωρίζετε ε, τη γεωγραφική περιοχή της εντολής μου. Ε, έτσι όπως το βλέπω εγώ και οι συνάδελφοί μου και στην ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης και πρέπει να ξεχωρίσουμε τρία επίπεδα. Έχουμε μία σειρά χωρών, υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των χωρών και υπάρχει και η θέση της περιοχής σε ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο. Όλα αυτά αλληλοτροφοδοτούνται. Οι προκλήσεις τώρα. Είναι πάρα πολύ εύθραυστη η περιοχή αυτή ε, προς νότον μιας άλλης ευαίσθητης περιοχής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα λοιπόν είναι αλληλένδετα και αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Θα είμαι πολύ ειλικρινής. Ε, αν δεν προσέξουμε αυτή την περιοχή ε, θα ε, μας, θα, θα, θα, θα μας έρθει μπούμεραγκ. είναι μια περιοχή που έχει πάνω από 200 εκατομμύρια ανθρώπους. Τα θέματα διακυβέρνησης, το άνοιγμα της ε, κοινωνίας σε ένα επίπεδο είναι η μεγάλη πρόκληση και αυτό το λέω γιατί πάω πέρα από τον κλασικό εκδημοκρατισμό και τις σωστές εκλογές. Το θέμα είναι αυτή η περιοχή αναπτύσσει θεσμούς που θα μπορέσουν να απορροφήσουν ε, το σεισμικό αποτέλεσμα ε, των διαφοροποιήσεων Καμιά φορά ναι, σε κάποιες χώρες ναι, σε άλλες χώρες υπάρχει στασιμότητα. Και αν δείτε το Νότιο Σουδάν για παράδειγμα, η κατάσταση είναι καταστροφική και σε ανθρώπινο επίπεδο και σε θεσμικό και σε επίπεδο συνόρων και, και στο ευρύτερο πολιτικό ζήτημα. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι και γι' αυτό χαίρομαι που είμαι μαζί σας, γιατί είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση. Υπάρχουν και εσωτερικές πιέσεις τώρα και υπάρχει και ο αντίκτυπος, η επίδραση νέων εξωτερικών επιδράσεων στην περιοχή. Δηλαδή τα παρεπόμενα, ε, οι παρεπόμενες επιδράσεις της ε, σύγκρουσης στον κόλπο. Θα επανέλθω σε αυτό, αλλά να το έχετε υπόψη σας. Υπάρχει δηλαδή αυτή η συνεχής ροή επιρροών και αντίθετων επιρροών. Τα προβλήματα στην περιοχή είναι η οικονομία, δηλαδή εμείς έχουμε μια δημογραφική έκρηξη και είναι ένα ερώτημα αν η οικονομική ανάπτυξη, για να μην μιλήσουμε για τη διαχείριση της αναδιανομής των ωφελών από το, την ανάπτυξη, θα φτάσουν σε αυτό τον πληθυσμό που ολοένα ε, ε, αυξάνεται. Είναι μια, ε, ένα μαθηματικό πρόβλημα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν είναι ωφελούμενοι από αυτή τη διαδικασία, αναπόφευκτα θα κάνουν ένα από τα δύο είτε θα μεταναστεύσουν ε, μέσα στο μυαλό τους, δηλαδή δεν είναι πια αφοσιωμένοι στο κράτος. Το κράτος δεν μπορεί να είναι η τελευταία καταφυγή για να ε, εξασφαλίσει την αφοσίωση των πολιτών που έχει να κάνει αυτό με την πολιτική διαχείριση ή κακοδιαχείριση ή φεύγουν κανονικά. και επειδή δεν μπορούν να πάνε στο νότιο Σουδάν, δεν είναι καλό μέρος αυτό, πάνε προς τα βόρεια. Δεν το λέω για να σας ανησυχήσω, απλώς πρέπει να δούμε πολύ ρεαλιστικά την κατάσταση. Και δεν μπορούμε να λέμε μόνο κοινοτυπίες και ε, η πολιτική μας να είναι η δημιουργία μικρών χωριών. Ε, Εμεί κάναμε πολύ σοβαρή δουλειά για το θέμα αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι να ξέρουμε την τάξη μεγέθους του προβλήματος με την πολιτική διαχείριση και είτε μιλάμε για την Ερυθρέα, Αιθιοπία, Σομαλία, Σουδάν, Νότιο Σουδάν, Τσιμπουτή, Κένια και την Ουγκάντα ε, αυτές οι δύο τελευταίες ε, ε, δεν είναι στο, στο κέραστο καθ' αυτά. Η διαχείριση λοιπόν είναι μη ικανοποιητική και είναι αμφισβητή συζητήσιμες οι πολιτικές επιλογές και η πολιτική διαχείριση. Βέβαια, εύκολα μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποια καθεστώτα, αλλά το θέμα είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εδώ, γιατί είναι προς το συμφέρον μας επίσης. Γι' αυτό είπα ότι η δημοκρατία καθ' αυτή θα πρέπει να στηρίζεται σε τέτοια περιοχή ε, σε μια πολιτική κατανόηση και θεσμική δυνατότητα πλουραλισμού που θα μπορεί να διαχειρίζεται τις διαφορές δηλαδή είτε είναι εθνοτικές είτε θρησκευτικέ είτε οτιδήποτε. Αν δεν υπάρχει αυτή η βάση τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό το είδαμε και στη Σομαλία και στο Σουδάν και στο Νότιο Σουδάν με τρόπο πραγματικά ε, καταστροφικό σε ό,τι αφορά την τάξη μεγέθους και αυτό θα μας πάει σε θέματα ασφάλειας αργότερα. Τώρα, το μεγάλο θέμα που θέλω να θίξω, γιατί σας έδωσα μια ιδέα ε, σχετικά με το τι μεταβολές υπάρχουν στην περιοχή αυτή. Εφιστώ την προσοχή σας τις εξελίξεις στον κόλπο. Και εδώ θα ε, βάλω το θέμα σε πολύ ευρύτερο πλαίσιο και θα πρέπει να σκεφτείτε όλοι γεωστρατηγικά. Αυτή η περιοχή ε, ε, ε, είναι η ανατολική ακτή της Αφρικής πάει μέχρι την Ερυθρά θάλασσα και την Αίγυπτο. Είναι 30 με 40 χιλιόμετρα από την Ιεμένη, η απόσταση από την Ιεμένη και αυτά που γίνονται στην Ερυθρά θάλασσα. Εδώ το εμπόριο, ο πολιτισμός, και οι πολιτικές διασυνδέσεις ε, προϋπήρχαν πριν από την έλευση του πρώτου Ευρωπαίου. Ε, εμείς είμαστε οι πρόσφατοι αφιχθέντες εκεί. Τώρα όμως βλέπουμε την ανάδυση εκ νέου παλαιών συμφερόντων. Αυτό συμβαίνει στον κόλπο. Κάποιοι Αφρικανοί ομόλο, συνομιλητές μου ε, ε μιλούν για τις, ε, την, την εκμετάλλευση στην Αφρική που δεν θα είναι όμως εκμετάλλευση από τους λευκούς. Θα πρέπει να δούμε. Ε, οι, οι, οι χώρες αυτές ξέρουν ότι έχουν στο πολιτικό σύστημα. Πώς θα τα αντιμετωπίσουν και τι παίζεται εκεί αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως το βλέπω, μέσα από το πρίσμα της δικιάς μου εντολής στην περιοχή, είναι ότι πριν από την τελευταία ε, διένεξη με το Κατάρ των χρόνων αυτών, από την Ιεμένη τα τελευταία 5-6 χρόνια υπήρχε αυξανόμενο ενδιαφέρον ε, στο να εξασφαλιστεί η ασφάλεια ε, στη δυτική όχθη του κόλπου. Αυτό πιστεύουν στις χώρες του κόλπου και έτσι μου το εξήγησαν. Δεν έχουμε εμείς το μονοπόλιο ως Ευρώπη στην πολιτική γειτονία, έχουν και εκείνοι. Το θέμα είναι ε, μπορούμε να μην έχουμε παράλληλες σχέσεις αλλά μια συνεργασία η οποία ε, θα ε, καλύπτει την περιοχή ολόκληρη. Αυτό είναι το θέμα γιατί αλλιώς ε, διατρέχουν κινδυνό οι επενδύσεις μας και τα ενδιαφέροντά μας στο κέρας της Αφρικής. Μπορούμε να εντάξουμε και το κέρας της Αφρικής σε όλη αυτή την εικόνα. Τώρα, ένα θέμα είναι ότι οι χώρες αυτές νιώθουν ότι υπάρχουν, ε, αντιμετωπίζουν πιέσεις για να ε, προσχωρήσουν σε μια συμμαχία. Δεν είναι πρώτη φορά αυτό. Πολλοί από μας ε, προερχόμαστε από χώρες ε, που ε, αντιμετώπισαν αυτές τις πιέσεις να ενταχθούν σε συμμαχίες και αυτές οι χώρες στην Ανατολική Αφρική και το κέρας της Αφρικής αντιμετωπίζουν και αυτές τέτοιες πιέσεις. Το θέμα που πρέπει να λύσουν είναι το εξής. Θα πάρουν το μέρος κάποιου, θα ταχθούν υπέρ μιας πλευράς έτσι το βλέπουν, και τι κόστος ε, εσωτερικής ισορροπίας θα πληρώσουν. Μην ξεχνάμε ότι αυτές είναι ή ως επιτοπλίστων μουσουλμανικές ή έχουν ανάμεικτο πληθυσμό και κοινότητες μουσουλμανικές και μη μουσουλμανικές. Και εκεί υπάρχουν δυνητικά ε, πολλές ε, διενέξεις που μπορεί να επιδεινωθούν ανάλογα με τις συμμαχίες που θα επιλεγούν. Υπάρχει και ε, ένα ε, άλλο θέμα, ε, ο πειρασμός των χρημάτων. Κάποιος μου το είπε. Εμεί είμαστε φτωχοί, άμα μας δώσουν πολλά χρήματα τι θα κάνουμε. Δηλαδή το θέμα είναι πόσο φτηνά θα πουλήσει κανείς τον εαυτό του. Τουλάχιστον εγώ έκανα μια παρόμοια συζήτηση με δύο-τρεις ε, αρχηγούς κρατών ε, το να υπάρχει ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν έχει την εντολή τη δική μου και αυτό είναι προ τιμήν σα που το κάνατε. Για μερικά χρόνια ήταν προνόμιο να αισθάνομαι ότι άνθρωποι σημαντικοί στις χώρες αυτές, οι ηγέτες τους, ε, πιστεύουν ότι μπορεί να αποταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσουν συμβουλή σε πολιτικό επίπεδο. Δεν έχουν κανέναν άλλον συνομιλητή που αλλού να πάνε. Αυτό σημειώστε το και κρατήστε το γιατί είναι σημαντικό. Τώρα το αν αξιοποιείται όπως πρέπει, ε, ε, αυτό έχει να κάνει και με το δικό μου, τη δική μου ικανότητα και την ικανότητα των συνεργατών μου. Τώρα, εμείς είχαμε κάποιες εντάσεις λοιπόν που τροφοδοτούν φυγόκεντρες τάσεις και στο εσωτερικό των χωρών και στο εσωτερικό μιας περιφέρειας. Υπάρχουν λοιπόν φυγόκεντρες δυνάμεις. Πώς θα τις κρατήσουμε τις δυνάμεις εκεί. Άμεσα η πρώτη αντίδραση είναι συνομιλήστε. Ε, υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη που μου ζήτησαν να πάω, με καλούν και από εκεί. Απαντώ όμως, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι η λύση, διότι θα πρέπει η περιοχή αυτή να αρχίσει να σκέπτεται πώς θα διαχειριστεί ε, καλύτερα, τον, ε, πώς θα διαχειριστεί τα του οίκου της και πώς θα συνεργαστεί με άλλους. Πιο συγκεκριμένα, η Σομαλία, μια χώρα που ε, στη, χάρη στην υποστήριξή σας ε, που σημαίνει επενδύσεις στην ασφάλεια, αναπτυξιακά έργα κλπ. Χάρη σε όλα αυτά γυρίζει σελίδα η Σομαλία, αλλά επουδενή δεν έχει φτάσει σε ασφαλή λιμένα. Τώρα θα πρέπει να πορευτεί μέσα σε θύελα γιατί ξαφνικά βλέπουν ότι πιέζονται να πάρουν μέρος, να πάρουν θέση σε μια σύγκρουση που δεν θεωρούν ότι είναι δική τους η σύγκρουση αυτή, αλλά πρέπει να επιλέξουν. Αυτό είναι σημαντικό. Και εμείς έχουμε ζωτικό ενδιαφέρον να φροντίσουμε ώστε το, να μην ε, ε, πάει προς λάθος κατεύθυνση η Σομαλία. Τώρα περνάει από μια θύελα πολιτική η χώρα και πρέπει να δοθεί κάθε βοήθεια. Η Ερυθρέα. Η Ερυθρέα έκανε την επιλογή της. Ήδη ε, έφτασε ένα λιμάνι. Η Ερυθρέα είναι δύσκολη, δύσκολο να κατανοηθεί. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Η Αιθιοπία αντιμετωπίζει τα θέματα, είναι αρκετά μεγάλη για να τα καταφέρνει σε ένα μεγάλο βαθμό. Το Σουδάν επίσης έχει διασυνδέσεις ε, με πολλές χώρες του, κόλπου. Το Τζιμπουτί, όπως είπε ο πρόεδρος, έχει πάρει θέση, αλλά ε, κρατάει και λεπτές ισορροπίες. Ε, το Σομάλιλαντ που είναι μέρος της Σομαλίας αλλά δρά ανεξάρτητα για να το πω έτσι έχει σαφώς πάει με το μέρος της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, επεξεργαζόμεθα το τι μπορεί να συμβεί. Εδώ θα σας πω τα βασικά. Η ανατολική ακτή της Αφρικής, ε, ερυθρά και προς τα κάτω, ε, έχει στρατιωτικοποιηθεί σε ε, βαθμό ανευπροηγουμένου. Δηλαδή η δυτική πλευρά της ερυθράς θάλασσας έχει ε, ενταχθεί σε μια στρατιωτική κρίση η οποία εκτιλήσεται στον κόλπο, στην Ιεμένη. Και έχουμε διεθνοποίηση της κρίσης ασφάλειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ένα λιμάνι μετά το άλλο ε, μισθώνεται, ε, αποκτάται και αποκτά στρατιωτική βάση. Ποιες είναι οι επιπτώσεις όλων αυτών. Θέτω τα ερωτήματα, αλλά δεν έχω τις απαντήσεις. Πάντως ε, είναι γεγονός ότι υπάρχει στρατιωτικοποίηση. Και αυτό σε μια εποχή όπου πολλές από αυτές τις χώρες χρειάζονται απελπισμένα πιο πολλές επενδύσεις. Τι επενδύσεις και με ποιους όρους. Ε, θα υπάρξει ανταγωνισμός για να ε, βρεθούν συνασπισμοί και πάλι ε, για να, να υπάρξουν συμμαχίες και συνασπισμοί τι κόστος πρέπει να καταβληθεί. Τα τελευταία 25 χρόνια τέλος και αυτό είναι από τις επιτυχέστερες περιπτώσεις προσιλητισμού που είδαμε ε, εδώ και πολλές δεκαετίες, δηλαδή την έλευση του Ουαχάμπη σαλαφισμού σε αυτή την περιοχή. Αυτό γιατί το θέτω, γιατί τολμώ να θέσω αυτό το θέμα ως μη μουσουλμάνος εγώ. Ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή που είναι γνωστή για τη διαφορετικότητα των πληθυσμών, της, της ιστορίας και επειδή υπάρχει εκεί ανάγκη συνύπαρξη, συνύπαρξης, η ε, εμφάνιση μιας πίστης ε, ενός δόγματος που αρχίζει να ε, κάνει κάτι που είναι άνευ στην αποκλειστικότητά του. Μιλάω για μια διάβρωση των δυνατοτήτων συνύπαρξης. Η αφοσίωση, η ταυτότητα αρχίζουν να αλλάζουν. Δεν ε, περιμένετε να, από μένα να σας πω πού μπορεί να οδηγήσουν όλα αυτά. Αλλά το θέμα υπάρχει, είναι πραγματικό. Ε, πολλοί το αντιμετωπίζουν με ευγενικά, το περιγράφουν με εφημισμούς, μιλάνε για βίο, εξτρεμισμό κλπ. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει ρίζοσπαστικοποίηση ε, των πληθυσμών που αρχίζουν να λένε ότι η αφοσίωσή τους ε, είναι προς κάτι άλλο από το μεταπικιακό κράτος αυτής της περιοχής της Αφρικής. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Ε, το έχω συζητήσει και με ηγέτες εκεί και σε όλα τα επίπεδα των, της κοινωνίας έχω κάνει συζητήσεις και βλέπω ότι υπάρχει μία ε, αυξανόμενη ανησυχία ή η οποία ανάγεται αν θέλετε και σε θέματα πολιτικής οικονομίας γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ότι συνεχώς ε, υπάρχει ροή κεφαλαίων ε, ε, προς τα έξω. Η ριζοσπαστικοποίηση γίνεται αυτόνομη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε. Και ξαναγυρίζω στο θεμελιώδες ερώτημα. Έχουμε ε, την πρακτική και τους θεσμούς του πλουραλισμού πριν μας απασχολήσει το ε, ένας ε, πολίτης μία ψήφος. Σήμερα έτσι όπως είναι τα πράγματα μπορεί μία γυναίκα να μην έχει μεγάλες ευκαιρίες. Αν συνδυάσουμε τα τρία αυτά στοιχεία θα πρέπει να δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε. Ποιες είναι οι προκλήσεις που συζητώ εξ ονόματός σας με τους συνομιλητές μου στην περιοχή. Πρώτον, η Ερυθρά. Η Ερυθρά θάλασσα τώρα έχει γίνει μεγάλο θέμα. Τι σημαίνει για μας στην Ευρώπη. Μία, μία ασφαλής στρατιωτικοποιημένη ε, ερυθρά θάλασσα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο 60% του εμπορίου μας. Αυτό είναι το θέμα και χαίρομαι που οι Αφρικανοί ε, συνομιλητές μου το καταλαβαίνουν αυτό γιατί θίγονται και εκείνοι. Μετά, ο Νίλος ε, η άλλη μεγάλη υδάτινη αρτηρία που έγινε αντικείμενο διαφοράς μεταξύ Αιθιοπίας, Σουδάν, Αιγύπτου και όλο και προς τα κάτω. Ε, λόγω της σημερινής κατάστασης στον κόλπο ε, βλέπουμε πολλή δραστηριότητα γύρω από τον Ήλο, από την Αίγυπτο, που ανησυχούν για τη διαχείριση των υδάτων του Νείλου, αλλά υπάρχει και ένα θέμα με τα νερά προς τις πηγές, όπου και εκεί ε, υπάρχουν αξιώσεις ε, διαχείρισης των υδάτων. Τέλος η μετανάστευση. Ενώ εμείς ανησυχούμε για τη μετανάστευση προς την Ευρώπη, υπάρχει μετανάστευση η οποία γίνεται συνεχώς και σε τεράστια κλίμακα στην Αφρική, από χώρα σε χώρα. Και <clears throat> πηγαίνουν σε αφιλόξενες περιοχές με μεγάλες δυσκολίες, εμείς δίνουμε πολλά χρήματα πολύ σωστά για διάφορους λόγους, δηλαδή και ανθρωπιστικούς και για καθαρά συμφεροντολογικούς λόγους. Τα κάνουμε αυτά. Συμβαίνουν. Αν δείτε όμως ε, τις δημογραφικές αλλαγές, ε, εγώ τουλάχιστον βλέπω ότι υπάρχει ένα φράγμα το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει. Ε, ο αριθμός των ανθρώπων που μπαίνουν στην αγορά εργασίας κάθε μέρα ξεπερνάει κατά πολύ την οικονομική δυνατότητα απορρόφησής τους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι πρέπει να κάνουμε και με ποιον άλλον θα συνεργαστούμε. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Επίσης, τα σύνορα στην περιοχή αυτή, τα απικιακά σύνορα δεν είναι τελεσίδικα. Ε, θα πρέπει να υπάρξει οριοθέτηση. Επίσης υπάρχουν φυσικοί πόροι και εκεί βρίσκονται ομάδες ανθρώπων που είναι περιθωριοποιημένες. Το θέμα είναι πολιτικό και εμείς έχουμε να παίξουμε μεγάλο ρόλο γιατί ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία. Ένας Θεός ξέρει πόσο εμπειρία έχουμε από τη δημιουργία συνόρων που μπορούν να τύχουν καλύτερης διαχείρισης. Μίλησα για τη ριζοσπαστικοποίηση. Και για να κλείσω, θέλω να πω ότι δεν θέλω να έρθω εδώ και να σας δώσω την εντύπωση ότι βαράμε το καμπανάκι του κινδύνου και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Πρώτος κανόνας, το λέω και το ξαναλέω και στους συναδέλφους μου, δεν πληρωνόμαστε για να είμαστε θεατές. Μας πληρώνουν για να εκπροσωπούμε συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διακυβεύονται. Πώς θα τα προασπίσουμε, με ποιο τρόπο, πώς θα θέσουμε προτεραιότητες. Πρώτον, λόγω της εσωτερικής διαφωνίας που έχουμε σε ορισμένες χώρες είναι ζωτικό να παραμείνουμε στις θέσεις μας και να δούμε αν μπορούμε να προωθήσουμε την συμφιλίωση, τη συνδιαλλαγή. Γιατί αν το σοφράγμα σπάσει σε αυτές τις χώρες, τότε θα υπάρξει υπερχείληση και θα αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα. Το Νότιο Σουδάν είναι το μεγάλο παράδειγμα. Εδώ ήταν παλιά η Σομαλία πριν από 10 χρόνια. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Ε, πρέπει να, εστιάσουμε, να είμαστε εστιασμένοι. Επίσης, ε, να δούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί, να οικοδομηθεί περιφερειακή ε, ολοκλήρωση. Η περιοχή καταλαβαίνει τώρα ότι αν δεν ε, προχωρήσει την ολοκλήρωση και τη συνεργασία, τότε θα διαμελιστεί θα γίνει ένα πτώμα ε, όπου τα όρνεα θα, θα αποκόβουν κομμάτια. Το ξέρουν αυτό. Θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε να αποτραπεί αυτό. Και έχουμε εμπειρία εδώ και από τη δική μας την ιστορία και από την εμπειρία της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να, να αλλάξουμε ε, αυτό το διάλογο κουφών σε κάτι πιο επικοδομητικό μεταξύ του κόλπου και της ε, περιοχής αυτής ούτως ώστε να έχουμε μια πιο παραγωγική σχέση. Και εδώ μπορεί να παίξουμε ρόλο. Σίγουρα εμείς ε, το ε, ξεκαθαρίζουμε αυτό προς πάσα κατεύθυνση, ότι δηλαδή είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Σταματώ εδώ, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Άλεξ. Ήταν πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Ε, νομίζω ότι αναφέρθηκε σε μια περιοχή ε, όπου υπάρχουν πολλές και διάφορες προκλήσεις και μας τα εξήγησε πολύ καλά. Έχουμε περίπου μισή ώρα μπροστά μας. Ε, θα δώσω το λόγο στον πρώτο μιλτή από το ΕΛΚ, ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είστε εδώ, είστε εδώ και πάλι μαζί μας κύριε Ρόντος. Ε, είναι πάντα διαφορετικά αυτά που μας λέτε. Σε σχέση με την προηγούμενη παρουσία σας, με τις προηγούμενες παρουσίες σας μάλλον, είχα την εντύπωση, δεν ξέρω αν είναι φιλοσοφικό ή έχει να κάνει με τον αριθμό των προβλημάτων και των προκλήσεων, αλλά έχω την εντύπωση περιπτώσει ότι έχει αλλάξει κάπως και εσεί την προσέγγισή σα. Είναι σημαντικό αυτό που μας υπενθυμίσατε, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου τη σημασία αυτής της περιοχής διότι βεβαίως εμείς εξετάζουμε τι γίνεται ε, στην άμεση γειτον, γειτονιά μας ανατολικά και νότια αλλά έχουν αντίκτυπο σε μας και γείτονες των γειτόνων μας και ίσως να το αγνοούμε αυτό καλό είναι που μας τα επενθυμίσατε. Επίσης θέλω να ξέρω τι εννοείται πιο συγκεκριμένα. Αναφερθήκατε στην ε, στρατικοποίηση της, κόκκινη της ερυθρής θάλασσας ε, ε, λιμάνι με το λιμάνι. Ποιος το κάνει αυτό όμως, ε, τα εν λόγω κράτη ή αναγκάζει το καθένας να πάρει θέση, για λεξη στρατόπεδο. πρέπει κάποιος να υποδεχθεί, να, να δεχθεί ε, ξένες ε, δυνάμεις στρατιωτικές. Ήταν λίγο ασαφές έτσι όπως μας το είπατε. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε, να μας πείτε. Στο Πότ Σουντάν ε, συμβαίνει το τάδε, στο Τζιμπουτί συμβαίνει το Δίνα, στη Σομαλία, στο αεροδρόμιο, στο Μογκαντήσιο, το άλλο. Καλό είναι να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πού και ποιος ζητάει τι από ποιον. Θέλετε να απαντήσετε άμεσα ε, όπως θέλετε. Έχουμε χρόνο. Ίσως να μπορείτε να απαντήσετε τώρα, απευθείας. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που έχουν ερωτήματα. Ναι, ακούστε. Ναι, ίσως να είμαι λίγο, να το φιλοσοφώ πιο πολύ το πράγμα. Γι' αυτό ενδεχομένως να έχω να και τα μαλλιά μου. Ε, υπάρχει και η θρησκεία της οικονομίας. Σε πάση περιπτώσει, για τη Μασάουα τα πράγματα δεν είναι σαφή, αλλά σίγουρα ενδιαφέρονται τα Εμμυράτα για το Πόρτ Σουντάν στο, στο βορρά παραμένει υποσουδανική ε, κυριαρχία, αλλά γίνονται συζητήσεις ό,τι αφορά την Άσα, Νότια Ερυθρέα, μόλις πάνω από το Τζιμπούτι. Αυτό το έχουν πλέον τα Αραβικά Εμμυράτα ως στρατιωτική βάση, είναι επιχειρησιακή βάση, δηλαδή για την Ιεμένη, τον Τζιμπουτί τώρα. Εκεί βρίσκονται όλοι στο Τζιμπουτί. Τα οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Γαλλία, όμως κυρίω αυτό που έχει σημασία είναι η άφηξη της Κίνας με μια τεράστια επένδυση. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε ε, τελικά ποια είναι τα σχέδια και οι προθέσεις της Κίνας. Αλλά πάντως η, επένδυση είναι τεράστια. Το ίδιο ισχύει και για τη Σαουδική Αραβία, έχει και αυτή η βάση. Μετά έχουμε στη Σομαλία την Μπέρμπυρα, εκεί βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γίνεται μια συζήτηση είναι μια στρατιωτική βάση που θα συνδεθεί με το λιμάνι, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος θα την επανδρώσει. Τώρα, στο λιμάνι του Μποσάσου, και αυτό ε, ελέγχεται από συμφέροντα των Εμμυράτων. Το Μογκαντήσιο είναι στα χέρια της Τουρκίας. Οι Τούρκοι το ε, διαχειρίζονται. Πιο κάτω, σε ό,τι το Κισμάιο, ακόμα δεν το έχει αναλάβει κάποιος, όμως να βάλουν χώρα συζητήσεις, πάλι με συμφέροντα των Εμμυράτων. Ε, λοιπόν, είναι ένα στοιχείο είναι ένα παιχνίδι εμπορικό το οποίο όμως πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε στρατιωτικό παιχνίδι λόγω της συγκυρίας. Δηλαδή το στρατιωτικό σκέλος ε, πήρε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη διαστάσεις. Επίσης όταν τα αναφέρω αυτά πρέπει να ξέρω ότι όταν έχουμε μια χώρα σαν την Αιθιοπία 100 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα και παρακολουθούν πολύ προσεκτικά διότι ε, το Τζιμπουτί είναι η μόνη έξοδος για αυτούς ε, προς τη θάλασσα. Έτσι λοιπόν για την Αιθιοπία είναι πολύ σημαντικό ζήτημα ασφάλεια αυτό. Ε, γι' αυτό λοιπόν αναφέρομαι στη διεθνοποίηση του, προγράμματος, του, του προβλήματος της ασφάλειας. Ελπίζω να σας έδωσα κάποια στοιχεία, κάποια περαιτέρω στοιχεία. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο κ. Παντζέρη τώρα έχει το λόγο για το S&D. Ευχαριστώ πολύ. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, εισαγωγική σας έκθεση. Πολλά πράγματα θα μπορούσα να πω, αλλά θα ήθελα απλώς να κάνω κάποιες ε, σύντομες παρατηρήσεις σε σχέση, ερωτήσεις μάλλον, σε σχέση με αυτά που λέγατε. Πρόκειται για μια ασταθή περιφέρεια. Πέστε μου, στην ουσία οι εξωτερικοί ή οι εσωτερικοί παράγοντες σταθερότητας παίζουν μεγαλύτερο ρόλο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία τα οποία έχουν χαρακτηρίσει την πρόσφατη ιστορία της ε, ε, ε, περιοχής, τις αναφέρατε και εσείς, αναφέρατε και εσείς τις διάφορες ε, δυνάμεις της περιοχής, τα στοιχεία της παγκόσμιας οικονομίας, τις τοπικές σειράξεις, τον ρόλο των εξωτερικών δυνάμεων και των αναδειωμένων παραδοσιακών δυνάμεων. Κάνω την παρατήρηση αυτή γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να ξέρουμε επί ποιων στοιχείων συζητούμε γιατί λέμε ε, ποιοι είναι οι παράγοντες σταθερότητα, Αλλάζει το παιχνίδι αν οι παράγοντες είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί. Δεύτερη παρατήρηση. Αναφερθήκατε ή μάλλον ε, ε, ε, θέσατε ένα ρητορικό ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχουμε κάποιες δυσκολίες παρέμβασης που οφείλονται στο γεγονός ότι έχουμε πρόβλημα να καθορίσουμε κάποια ε, πρόγραμμα παρέμβασης ή γιατί τα ε, ε, συμφέροντα είναι διαφοροποιημένα και επομένως δεν επιτρέπουν μια κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, αναφερθήκατε στη στρατιωτική βάση που έχει πλέον η Κίνα ε, εδώ και λίγο καιρό. Η Κίνα είναι ένα πρόβλημα. Ε, τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, τα όσα συμβαίνουν ε, λόγω της μετανάστευσης θα πρέπει να μας οδηγήσουν να συζητήσουμε, να θέσουμε επιτάπητος κάποια προβλήματα γιατί υπάρχουν γόνες, ζώνες οι οποίες όπως ας πούμε του κέρατος της Αφρικής που είναι ιδιαίτερος ασταθής. Ε, θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποια, ποιος είναι ο ρόλος, ακριβώς τι κάνει αυτή η μεγάλη δύναμη ε, στην Αφρικανική Ήπειρο. Άλεξ, έχει το λόγο. Ναι, δεν αφορά μόνο εμάς ε, και πραγματικά θα ήταν λάθος να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι και προσπαθούμε να λύσουμε τα ζητήματα αυτά. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν άμεσα θέματα στην περιοχή. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι η διεθνής κοινότητα με την ευρία έννοια ε, αυτή τη στιγμή ε, έχει στρέψει την προσοχή της αλλού. Από διατλαντικής πλευράς ε, τα πράγματα είναι πολύ συγκεχημένα. Δεν ξέρουμε ποια είναι η κατεύθυνση τελικά που ακολουθούμε. Και ούτε στην περιοχή αυτή είναι σαφές, σαφής οι προθέσεις των Αμερικανών, των ΗΠΑ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ο κόλπος δεν είναι μία ενότητα, οι χώρες του κόλπου με τις οποίες μπορούμε να συνοηθούμε, είναι αυτή τη στιγμή διαιρεμένοι, διχασμένοι. Μετά είναι η Κίνα. Ε, συμφωνώ πολύ τα μαζί πρέπει να μιλήσουμε με την Κίνα. Ακόμα και αν κάποιες συζητήσεις ε, οδηγήσουν σε απόκληση απόψεων σε διαφωνία, ας τα συζητήσουμε ότι ναι, πρέπει να πλώσουμε το δίκτυ μας ε, περισσότερο. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις, να ανοίξουμε δρόμους για τις μελλοντικές συζητήσεις. Βεβαίως αυτό που με ανησυχεί είναι ότι πρέπει να είμαστε πολιτικά αποτελεσματικοί στις συζητήσεις αυτές. Και για να είμαστε πολιτικά αποτελεσματικοί πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε. Ιδάλλως θα χαθούμε θα χαθούμε στις διαδικασίες ενώ η περιοχή θα καίγεται. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Οπότε συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά μην ξεχνάμε ότι, ξέρετε, οι άνθρωποι στρέφουν την προσοχή τους ε, προς ένα σημείο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Σε αυτήν την περιοχή, λόγω αυτών που σας περιέγραψα μόλις, θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σταθερά και απευθύνονται σε μας σε μια εποχή αβεβαιότητας. Αυτό είναι μία ακόμα πρόκληση και μία ακόμα ευθύνη για μας. Αλλά πρέπει σε αυτή την ευθύνη εμείς ε, να ανταποκριθούμε. Πάντως ε, ε, σημείωσα αυτό που μας είπατε. Μάλιστα, Τσάλς Τάνοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω Αλεξάνδρου. Έχει περάσει καιρός. Την τελευταία φορά μόλις είχες ε, ε, οριστεί, είχες διοριστεί ε, ω υπεύθυνο εκπρόσωπο προσωπικού για το κέρα τη Αφρική και κλείνουν και πέντε χρόνια από την έκθεσή μου. Ε, είχα καιρό να το διαβάσω, διαβάσω την έκθεσή μου πριν από λίγο την ξαναδιάβασα και διαπιστώνω ότι τα περισσότερα από αυτά που θεωρούσα τότε ε, ότι είναι σημαντικά και είχαμε υποβάλει και συστάσεις δεν έχουν επιληθεί. Ε, ο σαλαφισμός ε, των Βαχαμπίτων, ε, η φτώχεια, η πείνα. Συνάντησα τον Νίκολα Γκρουέσκι, τον Πρωθυπουργό της Μακεδονίας και μου έλεγε ότι φτάνουν οι βαχαμπιστές, οι φοχαμπίτες στη χώρα του. Η νεολαία ριζοπαστοκοποιείται. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και καιρό λοιπόν. Αυτό όμως που έχει αλλάξει επειδή αναφέρθηκε στον κόλπο ε, και στη μεγάλη αυτή, στο μεγάλο καυγά ε, με την μουσουλμανική αδελφότητα και το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία υπάρχει ένας διχασμός, υπάρχουν δικρόμενα συμφέροντα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο το οποίο δεν ανέφερε, είναι το θέμα του Brexit. Θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύει ότι θα γίνει με την επιχείρηση Αταλάντα, που είναι μια success, ένα success story για την καταπολέμηση τη πειρατεία ε, στι Ομαλικέ ακτέ. Ο προηγούμενο πρόεδρο τη Ομαλία ε, με ευχαρίστησε όταν το συνάντησα για την έκθεσή μου και γι' αυτό που έκαναν οι Βρετανοί και ο Βασιλικός στρατό είχα γράψει ένα έγγραφο και είχα πει ότι θα μπορούσε να εξακολουθήσει ε, να, το αρχηγείο να βρίσκεται στο μένα Βασίλειο ακόμα και μετά το Brexit αυτή τη επιχείρηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να σχολιάσετε από αυτό. Ε, τώρα για το θέμα της Σομαλίας. Ε, να πω ότι ένα από τους λόγους για τους οποίους ε, έχει ακολουθηθεί η γραμμή της Σαουδικής Αραβίας εκεί είναι επειδή θεωρούν ότι η Σαουδική Αραβία που αντιτίθεται περισσότερο ε, ε είναι σημαντική ανεξαρτησία για αυτούς και επειδή η Σαουδική Αραβία έχει μεγάλο ειδικό βάρος στην, ε, στον Αραβικό Σύνδεσμο ε, θα μπορούσαν κάποια στιγμή να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία τους είναι πάντως ένα σημείο σταθερότητας και μετριοπάθειας και κάποια στιγμή θα λάβουν την εξαρτησία τους. Δεν βλέπω δηλαδή πώς η Σομαλία μπορεί να ε, επανενωθεί. Αλλά υπάρχει βεβαίως ε, και εκεί και η πίνα πείνα. Πρέπει να δούμε πώς θα επιληθεί και αυτό το πρόβλημα. Επίσης θα ήθελα να ξέρω τι πρόοδος έχει σημειωθεί στην Ίγκαρ, σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση είχα κάνει κάποιες συστάσεις τότε σε ό,τι αφορά τις υποδομές, την οικονομική συνεργασία. Έχει συμβεί κάτι τα τελευταία πέντε χρόνια. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, διότι δεν γνωρίζω εγώ κάτι να έχει συμβεί. Βεβαίω υπάρχει και το λιμάνι του Μπέρμπερα, ανησυχώ για την στρατικοποίηση αυτού του λιμανιού και για τον Τζιμπουτί βλέπουμε ότι εμφανίζεται η Κίνα αλλά και η Ιαπωνία έχει εδώ και κάποια χρόνια βάση εκεί. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χειροτρέψουν τα πράγματα ε, στην Νοτιοανατολική Ασία με τους Κινέζους και τους Ιαπωνές να έχουν και οι δύο βάση πολύ κοντά η μία στη μία στην άλλη στη συγκεκριμένη περιοχή. Η επιχείρηση Αταλάντα ήταν πραγματικά εξαιρετική διαδικασία και νομίζω ότι πλέον ε, ε, αναφέρεται όχι μόνο στην πειρατεία, αλλά στη γενικότερη ασφάλεια των θαλασσών, στην θάλασσα του Έντεν και ε, σε όλη την περιοχή, ιδίω ανάμεσα στην Ιεμένη και την Σομαλία εκεί που κινείται άλλωστε και επίσης έχει να αντιμετωπίσει ε, και το παράνομο εμπόριο, κυρίως διακίνηση ναρκωτικών που προέρχεται από τον ε, ε, Ινδικό ωκεανό και πηγαίνει προς την Ανατολική Αφρική. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να διαβρύνουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την έννοια της θαλάσσιας ασφάλειας η Αταλάντη, πραγματικά η επιχείρηση Αταλάντα έδωσε την δυνατότητα να δούμε τα πράγματα ε, διαφορετικά και θα πρέπει να εστιάσουμε στα θέματα. Τώρα, το, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν ή θα επιλέξουν τα κράτη-μέλη να ε, χειριστούν το θέμα δεν το γνωρίζω, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και θα είναι πολύ αρνητικό εάν το αρνηθούμε. Το Σομάλιλαντ είχαμε ανταλλαγή απόψεων και για το θέμα αυτό στο παρελθόν δεν μπορώ να φανταστώ την ε, Σαουδική ε, Αραβία να υποστηρίζει την ε, απόσχηση. Ίσως να κάνω λάθος, αλλά πάντως έχω την εντύπωση ότι για την Σομαλίλανδη τα συμφέροντα είναι συγκεκριμένα και επομένως τον ε, Νίγηρα γίνεται πολλή συζήτηση σχετικά με το που θα πρέπει να επικεντρωθούν ε, τα ε, ζητήματα. Υπάρχουν και οι πρόσφατες εξελίξεις, γιατί εκεί είναι όντως θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να φέρουμε την πολιτική ολοκλήρωση, ενσωμάτωση της περιοχής και επίση να σας πω ότι μας βοήθησαν πολύ στη δημιουργία ε, των Federal States. Και όσο για το Τζιμπουτί έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά πώς μπορούν να πώς μπορούν αυτά τα διαφορετικά συμφέροντα που είναι παρόντα στο Τζιμπουτί να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να επιφέρουν ισορροπίες, δεν το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νάρτα από την ε, Άλντε. Και εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσω την εξαιρετική ε, εισήγηση που κάνατε. Είναι από τις εξαιρετικότερες που έχω ακούσει ε, για ένα θέμα τόσο περίπλοκο όσο του κέρατος ε, της Αφρικής. Συγχαρητήρια, ήταν εξαιρετικά σημαντική και ενδιαφέρουσα η παρουσία σας. Μια σειρά ερωτήσεων θα σας υποβάλω ο πρίγκιπας της Σαουδικής ε, Αραβίας, ε, η θέση του, το οικονομικό κόστος ε, που σημαίνει αυτό. Χοδιοκτισμός ε, λοιπόν του πρίγκιπα ε, ε, σε μια χώρα η οποία στην ουσία τρώει από τα αποθηκευμένα γιατί ξέρουμε ότι μειώνονται και τα αποθέματα πετρελαίου. Ε, επίσης το, το, το, το, η εγκληματική αυτή θέση κυρίως δε επειδή είναι και ε, σύμμαχος της Ευρώπης πώς, πόσο καιρό μπορεί να εξακολουθήσει να έχει τη στάση που έχει απέναντι και στην Ιεμένη ε, η Σαουδική Αραβία κατά την άποψή σας. Δεύτερον, συμφωνώ απολύτως. Το πρόβλημα της μετανάστευσης ε, ε, στην ουσία διαρκώς διονγκώνεται και επομένως θα πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν να δώσουμε λύσεις στους ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε θα πρέπει να υπάρχει μία δομή η οποία να μπορεί να καθορίσει ποια είναι ε, η ε, βοήθεια. Ε, η Αιθιοπία, ας πούμε, είναι σίγουρα μια χώρα η οποία μπορεί να επιβιώσει οικονομικά. Αλλά έχουμε την, το Νότιο Σουδάν, το οποίο πέρα από τον εμφύλιο πόλεμο ηγείται, έχει ηγεσία κλεπτοκρατική, ολιγαρχική, βασίζεται σε μια χώρα και σε ένα σύστημα φυλών. Στην περίπτωση του Βορείου Σουδάν επίσης έχουμε παρόμοια προβλήματα. Δηλαδή όπου και να γυρίσουμε να κοιτάξουμε δεν βλέπουμε να υπάρχει μια δομή η οποία θα μπορούσε να είναι αρμόδια για την ε, βοήθεια η οποία θα πρέπει να μοιραστεί στη χώρα, ε, στις χώρες. Ε, δηλαδή βλέποντας μια τέτοια ε, διευρυμένη διαφθορά δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα βοήθειας που θα ξεπερνάει βέβαια την απλή φιλανθρωπία. Τώρα, με μετά την ανεξαρτησία του του, του αυτοκράτορα Μενελίκ στην ουσία ξεχωρίστηκαν ε, ιστορικά ε, οι δύο περιφέρειες αυτές, ε, δηλαδή τη βόρεια από τη μία πλευρά και που φτάνει μέχρι τα βόρεια σύνορα της Κένιας και ξέρουμε ότι τα νότια σύνορα είναι τα αυτοκρατορικά σύνορα της ε, ε, Αιθιοπίας και η Σομαλία, ε, η οποία είναι η χώρα η οποία εθνοτικά είναι η πιο ενωμένη και η πιο ομοιογενής, στην ουσία είναι και αυτή που έχει τις περιοχές, είναι αυτή που έχει και τα μεγαλύτερα προβλήματα. από την άλλη πλευρά, το σημαντικό είναι ότι χάνεται το αξίωμα της εμπιστοσύνης προς την πολιτική αρχή και προς την κυβέρνηση. Όταν κανείς δεν έχει ούτε παρελθόν ούτε παρόν, τότε θα πρέπει να κοιτάξει μόνο προς το μέλλον, να δει τι υπάρχει παραπέρα. Um, well, uh, I think... Απάντηση. Νομίζω ότι μας δώσετε μία εικόνα ε, η οποία πραγματικά έδωσε κάποιες εξωτικές πινελιές στη δουλειά μου. Ε, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, δοκιχωτικές επινελιές έτσι στην ε, δουλειά μου και στη θέση που καλύπτω. Κοιτάξτε, εγώ μιλάμε για τους νέους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ανοιχτοί είναι οι νέοι, πόσο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το αφήσουμε. Η πολιτική της δικιάς μου γενιάς ε, στην ουσία δεν έχουν πια λόγο και θέση ε, σε αυτήν την ε, κοινωνία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να έρθουμε σε επαφή με αυτή τη νέα γενιά, με οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας, γιατί πραγματικά ενδιαφέρονται είναι και, και πολλοί θέλουν πραγματικά να κάνουν κάτι. Το ζήτημα δεν είναι ε, να τους πούμε ωραία λόγια, το ζήτημα είναι πώς μπορούν τα λόγια να γίνουν πράξεις. Ε, πρέπει να βελτιωθούν οι μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, να δημιουργηθούν θεσμοί οι οποίοι να έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν αυτούς, αυτούς τους νέους. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όλα τα άλλα που είπατε, η διαφθορά κτλ. Ναι, μα η νεολαία είναι ε, η πρώτη η οποία καταλαβαίνει ότι υποθηκεύεται το μέλλον της ακριβώς λόγω αυτής της ε, ε, ε, ε διαφθοράς. Κοιτάξτε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η μοίρα και το μέλλον της Σαουδικής Αραβίας. Με ενδιαφέρει περισσότερο η μοίρα και το μέλλον κάποιων άλλων ε, ε, χωρών που βρίσκονται απέναντι. Θα πρέπει να δούμε όμως πώς όλα αυτά τα λόγια, όλες αυτές οι ιδέες που έχουμε μπορούν να μεταφραστούν σε πράξεις, κυρίως δε πράξεις που να αφορούν τη νεολαία. Κάρβερ, Επιτίδιος και Αναγκόμες, οι τρεις τελευταίοι μας ε, ομιλητές. Ο Τζέιμς Κάρβερ που ξέρει τα πάντα για τη Σομάλιλαντ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονό ότι πάρα πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά ε, τα οποία ε, ακούσαμε και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε τα θέματα αυτά. Είναι σημαντική η περιοχή, το είπατε και, επίσης, και εσείς, το ξέρουμε ε, γενικά. Μας έχει, έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα της περιφέρειας αυτής ε, πολλές φορές ε, στην Επιτροπή μας ε, και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα. Ε, και το Κοινοβούλιο τουλάχιστον ενδιαφέρεται από πολύ στενά. Συμφωνώ με τα σχόλια ε, τα οποία κάνετε σχετικά με τη γεωγραφική σημασία και το γεωγραφικό βάρος. Ε, ναι, το κέρας της Αφρικής αντιμετωπίζει μια γενικευμένη κρίση, ναι, γιατί ξέρουμε ότι οι χώρες οι οποίες το αποτελούν αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα. Επίσης,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 Ήμουνα στην ε, Σομάλιλανδία ιδιωτική επίσκεψη ε, πέρσι και πραγματικά ε, εξεπλάγινε από τα στρατόπεδα των προσφύγων. Οι πρόσφυγες από την Ιεμένη έχουν ενταχθεί στη Σομαλική κοινωνία. Είναι ανοιχτή η Σομαλία απέναντι στους ανθρώπους αυτούς και αυτό με εξέπληξε. Λειτουργεί το σύστημα πολύ και γι' αυτό ακριβώς η Σομαλίλανδα αποτελεί και ένα πολύ καλό παράδειγμα. Επίσης αναφερθήκατε στην Σομαλία και τα ε, λιμάνια. Πρέπει να βρεθεί κάποια λύση εγώ δεν βλέπω την Σομαλία σαν project, εγώ την βλέπω ε, σαν μια ε, χώρα η οποία ε, μετά από 25 χρόνια προσπαθεί να βρει το, το δρόμο της ε, και η Σομαλίλανδ θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, δραχθεί, να δράξει τις ευκαιρίες έτσι ώστε να αναπτυχθεί. Αυτό που με ενδιαφέρει ε, είναι, είναι να υπάρξουν αυτές οι εξελίξεις. Βέβαια ακούμε για στρατηγικές που αφορούν συνολικά το κέρας, αλλά θα πρέπει να τις δούμε από κοντά. Δεύτερο σημείο Αναφερθήκατε σε διάφορα ε, λιμάνια, σε διάφορες ε, διαδικασίες. Ναι, το σημαντικό είναι να ε, υπάρχει και ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας που να τα συνδέει. Οι υποδομές λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ε, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με την ε, κυβέρνηση ε, έτσι ώστε να υπάρξουν συμφωνίες. Επίσης, ε, μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ριζοσπαστικοποίησης εάν δεν αντιμετωπίσουμε σωστά ε, την κοινωνία και τα ε, προβλήματά της. Υπάρχουν τμήματα της κοινωνίας τα οποία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι μόνο μέσω διεθνούς αναγνώρισης μπορεί η Σομάλιλαντ να προχωρήσει. Έχω χρόνο να μιλήσω ακόμα. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα η οικονομική ε, ε, ενίσχυση των εκλογών της ε, Σομάλια, των πολλών Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αφορά γενικότερα την ενοποίηση με την υπόλοιπη Σομαλία. Το θέμα είναι να δούμε εάν μπορούμε να παίξουμε κάποιο ρόλο στην προετοιμασία των εκλογών. Εάν ναι, είστε ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει number of questions on Okay. Um, to... Απάντηση. Δεν έχω χρόνο ε, δυστυχώς να απαντήσω διεξοδικά με τον τρόπο που θα έπρεπε να απαντηθούν τα ερωτήματά σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις, ε, ε οπουδήποτε απανταχού ε, τις δημοκρατικές, ε, συγγνώμη, εκλογικές ε, διαδικασίες αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αναγνωρίζουμε ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση όλες τις εκλογικές διαδικασίες, αλλά είμαστε υπέρ του ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο που πρέπει να υποθεί για τη Σομαλία. Η οικονομική, ε, η οικονομική υποστήριξη ε, εξισούται με αναγνώριση όχι. Ε, νομίζω ότι ε, καλύτερα θα ήταν να γίνουν, να επιταχυθούν οι εκλογές παρά το αντίθετο για να ξέρουμε ακριβώς ε, περί τίνος πρόκειται και τι, γίνεται ακριβώς. Γιατί τώρα όλοι αμφισβητούν την νομιμότητα των απαιτήσεων που η Σομάλιλαντ έχει για μεγαλύτερη αυτονομία, δημιουργία ανεξάρτητου κράτους κλπ έτσι προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το τι είναι αυτή η οντότητα, ποιο είναι το παιχνίδι που παίζει, περί τίνος ακριβώς ε, πρόκειται. Και αυτό είναι το κύριο ε, ερώτημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το δούμε με αυτό το τρόπο. Όσον αφορά τώρα το δυτικό, ε, ναι, το λιμάνι Μπαρμπάρι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, αλλά και όλα τα άλλα κράτη στην Σομαλία επίσης έχουν έρθει ε, σε μια συμφωνία και το ζήτημα εδώ είναι εάν μπορεί να προκύψει και κάποια συμφωνία με το Μογκαντήσιο. Να βρεθεί δηλαδή κάποιος τρόπος έτσι ώστε να δώσει κατά κάποιο τρόπο το πράσινο φως ε, στο ε, Κοινοβούλιο, γιατί έχουμε και Σομάλιλαντς που ε, είναι, εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Επιτίδιος. Ε, κύριε Ρόντο, σας καλωσορίζω και εγώ στην Επιτροπή και σας εύχομαι και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή. Ε, θα μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ και εγώ για την ε, εξαιρετική παρουσίαση και την γεωστρατηγική ανάλυση που μας κάνατε και πολύ σύντομα θέλω να σας ρωτήσω πρακτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μπορεί να συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής. Είπατε και ότι όλοι αναγνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, μία παράμετρο σταθερότητας. Και συμφωνώ με αυτό. Επαναλαμβάνω πρακτικά πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε αυτό. Δηλαδή, ποιες συγκεκριμένες ενέργειες πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να μπορέσει να αναμειχθεί θετικά στην όλη κατάσταση, όταν ξέρουμε ότι, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν αντιπαραθέσεις μεταξύ των ε, ε, κρατών, υπάρχουν εσωτερικές διαμάχες, υπάρχουν παρεμβάσεις ε, τρίτων δυνάμεων και, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ούτε κοινή εξωτερική πολιτική, ούτε στρατό, έχει μόνο χρήματα. Πώς λοιπόν πρακτικά μπορούμε ε, να παρέμβουμε ούτως ώστε να συμβάλλουμε στην ε, διαμόρφωση μιας θετικής ε, εξελίξεως στην περιοχή αυτή. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας πρώτα απ' όλα και ε, να σας απαντήσω αγγλικά. Um, what can the EU do? It's what the e already... Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ήδη κάνει πρέπει να είμαστε σαφείς. Υπάρχει μια τεράστια συνεισφορά, έτσι. Και δεν είναι μόνο χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει ιδιαίτερα στο να ακουστεί μία φωνή. Βοηθούμε δηλαδή την οικονομική ανάπτυξη, δίνουμε την οικονομική ελπίδα βεβαίως, ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των αντιμεχομένων. Να τους φέρει πιο κοντά, να τους φέρει στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν. Στη Σομαλία και αλλού. Γίνονται πολλά προς την κατεύθυνση αυτή. Τρίτον, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε περιφερειακές δομές. Και αυτό με πολλές δραστηριότητε. Εάν δηλαδή εσείς τώρα ρωτάτε, θέλετε να πείτε ότι δεν κάνουμε και τίποτα, όχι. Ε, γίνονται πολλά και μάλιστα αρκετά εντυπωσιακά. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα βεβαίως, πάντα. Όμως ρωτήθηκε προηγουμένως ε, κάτι σχετικό. Ήρθε η στιγμή πλέον να μην θεωρήσουμε ότι είμαστε οι μόνοι παίχτες. Πρέπει η στόχος μας να είναι να εμπλακούν και άλλοι. Έτσι ώστε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μοχλευθούν, αν θέλετε, μαζί με τα συμφέροντα άλλων για να μπορέσουμε όντως να σταθεροποιήσουμε αυτή την περιοχή. Να μην είναι απλά μια πηγή εξαγωγής προβλημάτων. Χρειαζόμαστε συμμαχίες στο εσωτερικό, στο εξωτερικό και είναι μια μακρά διαδικασία και δύσκολη. Εάν όμως συγκρίνουμε αυτή την κατάσταση τη σημερινή με αυτή που υπήρχε πριν από μερικά χρόνια στην περιοχή, μπορεί να πει κανείς ότι πάμε σωστή κατεύθυνση. Αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία που θα πρέπει να τονίσουμε. Και βεβαίω θα χρειαστούμε και τη δική σας βοήθεια, τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γι' αυτό. Να υπάρχει πίεση, να υπάρχει και ενθάρρυνση προς εμάς από την πλευρά σας. Τώρα κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να μην συμφωνήσουν, αλλά υπάρχει μια τάση ε, κάποια βαθιά πολιτικά προβλήματα να τα αναθέτουμε σε τεχνοκράτες. Εγώ προέρχομαι από μια σχολή σκέψης πολύ διαφορετική. Εγώ πιστεύω ότι άνθρωποι όπως εσείς πρέπει να δεσμεύονται περισσότερο και να συνεργάζονται και να εμπλέκονται για να βρεθούν λύσεις, για να έρθουν πιο κοντά αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολιτικό ζήτημα, είναι πολιτική πρέπει να μιλήσουν σε πολιτικούς. Με όλο το σεβασμό σε πολλούς από τους αδέλφους μου. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να σας ε, δώσω. Υπάρχει ένας ρόλος για σας. Τέλος, η Άννα Ναι, ευχαριστώ για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα αν και δραματική παρουσίαση των προκλήσεων των γεωστρατηγικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σε αυτή την περιοχή του κόσμου και ελπίζω αυτό να ξυπνήσει κάπως και τους ηγέτες μας διότι ως τώρα ε, δεν, δεν είχαν προνοήσει. Υπάρχουν βεβαίως γεωστρατηγικοί λόγοι, γεωπολιτικοί λόγοι που ε, μας οδηγούν τελικά στο να ε, παρακάμπτουμε ή στο να εθελοτυφλούμε απέναντι σε πολύ βασικά ζητήματα αρχών. Το Σουδάν δεν θα ήταν εκεί αν δεν είχαμε βοηθήσει στη δημιουργία του ακολουθώντας τους Αμερικανούς. Και μην ξεχνάμε βέβαια κάποιες κρίσιμες χώρες όπως η Αιθιοπία, όπως η Αίγυπτος. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς ε, μας προσλαμβάνουν ε, θεωρούν, θεωρείτε ότι έχουμε μια κοινή θέση, ε, ότι έχουμε κάποια θέση για την Ιεμένη παραδείγματος χάρη ή για την ε, ε αντι, αντι, αντιπαράθεση Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ ή εικόνα που δίνουμε είναι των εμπόρων όπλων ή μήπως είναι αυτή η εικόνα που δίνουμε είναι των εμπόρων όπλων. Μήπως είναι αυτή η εικόνα που δίνουμε στην περιοχή. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω ότι οι σχέσεις με τις χώρες αυτές συχνά είναι στα χέρια των ε, τεχνοκρατών και που μιλούν μόνο για ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν βλέπουμε δηλαδή πού βρίσκεται η αντίστοιχη πολιτική επιρροή που θα έπρεπε να υπάρχει με βάση τα, τις επενδύσεις, τις οικονομικές που έχουμε κάνει σε χώρες όπως η Αιθιοπία, ενώ θα μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά. Επιλέξαμε όμως να μην το κάνουμε. Ή επιλέξαμε να κάνουμε τη διαφορά για υπέρ των ε, καταπιεστών και όχι της νεολαίας που αναφερθήκατε κι εσείς και που θα καθορίσει το μέλλον της περιοχής και δεν έχουμε πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή. Η νεολαία ποια είναι. Θα την βρείτε στη, στη ζούγκλα του Καλέ. Θα δείτε εκατοντάδες αιθίωπες από την περιοχή. Και από την περιοχή αυτή, από την Αιθιοπία και από άλλες χώρες της περιοχής. Για να μην μιλήσουμε και για τις άλλες χώρες. Η Αίγυπτος τώρα. Ας είμαστε ειλικρινεί. Τι θα γίνει με την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Αυτοί δεν έχουν μαγευτεί από τα χρήματα των ε, Σαουδάραβων. Και σε αυτό το πλαίσιο, τι θα γίνει με τους Αμερικανούς. Είπατε ότι είναι σημαντικό το θέμα των ΗΠΑ. τι βλέπετε να συμβαίνει, προς τα πού πάνε οι Αμερικανοί. Θα ακολουθήσουν την οδό του Μπαράκ Ομπάμα που δεν ήταν και τόσο ευτυχής. Αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα. Άλεξ. Ναι, ευχαριστώ, Άννα. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, οι επιπτώσεις, ε, η εικόνα μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, έχει μια εικόνα η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Βεβαίως η εικόνα αυτή ποικίλει. Γενικά είναι μια εικόνα θετική. Ε, είναι, και το λέω αντικειμενικά αυτά είμαστε οι καλοί αν θέλετε, αλλά όταν είναι κάποιος καλός, ε, ορισμένε φορές μου θυμίζει την κριτική που είχε αναφέρει ο Ντένις Χίλι στο Βερονικό Κοινοβούλιο. Είναι, δεν είναι καλό να είναι κανείς πολύ καλός. Είναι σαν να μην έχουμε δόντια. Δεν, δεν ανησυχεί κανείς για τις επιπτώσεις δηλαδή αυτών που λέμε και αυτών που σκεφτόμαστε. Τώρα, θέσατε ένα πολύ καλό ερώτημα, το οποίο πρέπει όλοι να το έχουμε κατά νου. Η δική μου δουλειά είναι να υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να θεωρηθεί απλά ε, ένα ATM όπου κανείς τραβάει λεφτά. Ορισμένες φορές ε, μπορεί το ATM να μπλοκάρει την κάρτα. Αυτό ίσως είναι ένας τρόπος ε, να μετρήσει η άποψή μας. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχει λοιπόν μία βούληση ε, να ακουστεί αυτό που έχουμε να πούμε. Και βεβαίω κρατάτε και ποιες είναι οι ιδέες που έχουμε να προωθήσουμε. Δεν αρκεί να λέμε πρέπει να είστε καλοί με τους πολίτες σας Πρέπει να τους βοηθήσουμε να επιλύσουν ε, ζητήματα εσωτερική πολιτική που φαίνονται τελείως αδιέξοδα. Και αυτό που ήθελα να πω πριν πραγματικά για τους πολιτικούς, δεν το είπα για να σας κάνω κάποιο κομπλιμέντο ή για να σκολακέψω, αλλά για ασφαλιστικού λόγους. Τώρα για την Αίγυπτο και την Αιθιοπία είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και ιδιαίτερα τοξικό. Δεν ξέρω τι θα συμβεί τελικά. Αλλά είναι κάπως περίεργο. Δύο χώρες που θεωρητικά έχουν τα ίδια συμφέροντα. Έχουν τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους φόβους ενδεχομένως και παρεμφερείς δομές. Και παρόλα αυτά, εντάξει δεν έχει ξεκινήσει ε, κάποια εμπόλεμη κατάσταση, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Θα μπορούσε εύκολα να γίνει ένα τύχημα δηλαδή. Κάποιοι προσπαθούν διακριτικά να δουν πώς μπορούν να αρχίσουν κάποιες συζητήσεις. Υπάρχει περιθώριο να βρεθεί κοινό έδαφος. Και το πρώτο βήμα, κατά τη γνώμη μου, είναι και οι δύο χώρες να βοηθήσουν τον εαυτό τους και να μην εγκλωβίζονται στη γωνιά λόγω της δικής τους τριτορικής όπως έχει συμβεί τόσες φορές. Είναι δύσκολο κανείς να βγει από μια γωνία στην οποία έχει μπει ο ίδιος. Υπάρχει περιθώριο και υπάρχει κοινό έδαφος εφόσον φανούμε δημιουργικοί. Τώρα για τους Αμερικανούς. Ακούστε. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Ας είμαστε όμως προσεκτικοί, έτσι. Μη χαθούμε τώρα σε κάποιες καρικατούρες. Είναι μια μεγάλη χώρα, είναι ένα κράτος που λειτουργεί ως κράτος. Βεβαίω, ε, τα πρωτοσέλιδα είναι αυτά που ενδιαφέρουν σαν τους ε, ανθρώπους, αλλά υπάρχουν και πολιτικέ από πίσω. Υπάρχουν άνθρωποι με του οποίου συνεχίζουμε να μιλάμε. Και αυτή είναι η προσέγγιση που πρέπει να έχουμε. Ιδάλω ε, θα ε, απορροφηθούμε μόνο από αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση και στα πρωτοσέλιδα. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, δηλαδή, σε πολιτικό επίπεδο, διότι πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα προς όφελος ε, της συγκεκριμένης περιοχής. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι ε, αυτά τα 75 λεπτά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άλεξ που ήρθε στην Επιτροπή μας ε, για αυτή την παρουσίαση. Και νομίζω ότι αυτή η περιοχή θα πρέπει να μπει στην ατζέντα με το πρόγραμμα εργασιών μας για το 2018. Η Επιτροπή ΑΦΕΤ έχει προβλέψει μία επίσκεψη στην Αφρική το Δεκέμβριο, ίσως στην Αιθιοπία. Ο κ. Τάνοκ μας υπενθύμησε στην τελευταία έκθεση. Η τελευταία έκθεση ε, για αυτήν την περιοχή του κόσμου είναι, πάει, μας πάει ήδη πέντε χρόνια πίσω. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή τύχη στο έργο σας ε, κύριε Ρόντος. Θα κλείσει τώρα η συνάντησή μας. Αύριο το πρωί στις 9 θα συνεχίσουμε με τον Μάρκους Ίντερερ που θα είναι ο επόμενος πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μόσχα. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψε μαζί του. Καλό βράδυ σε όλους.